Buonasera a tutti. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους, όλους. Πάρα πολύ σύντομα και πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, να σας μεταφέρω αυτά που αποφασίσαμε σήμερα το πρωί στα πλαίσια της συνάντησης των ε, συντονιστών Έχετε ένα σημείωμα γύρω από τη συνάντηση αυτή, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταρχάς οι αποφάσεις που εκκρεμούσαν από την προηγούμενη συνάντηση, δηλαδή ο διορισμός των νέων μελών του ελεγκτικού, θα πρέπει σύντομα να οργανώσουμε τις ακροάσεις. Επίσης ο ορισμός της κυρίας Γκρέσλε για τη συμφωνία ο Ταυτόχρονα οι διαδικασίες σχετικά με τις ε, επιταχυμένες απλοποιημένες τελωνιακές ε, διαδικασίες, η έκθεση Λιμπεράσκη, σχετικά με την υπηρεσία, την εξωτερική, εξωτερική υπηρεσία. Ορίζουμε επίσης την κυρία Γκρέσλε αλλά περιμένουμε τις ενδείξεις από πλευράς της Επιτροπής σχετικά με το πακέτο τεσσάρων προτάσεων για την εξωτερική υπηρεσία, έτσι ώστε να διευκρινηθεί το ποιος θα κάνει τι, περιμένοντας επίσης και την υπόδειξη συντονιστού από πλευράς της σοσιαλιστικής ομάδας. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η συζήτηση για τον ορισμό του ενδιαμέσου προσωρινού Γενικού Διευθυντή της ΟΛΑΦ του κυρίου Άιλετ. Συζητήσαμε επί μακρόν παράλληλα και το θέμα της προκήρυξης για την κάλυψη ε, της θέσης, ε, της τακτικής πλέον θέσης ε, του Γενικού Διευθυντή της ΟΛΑΦ. Για το συγκεκριμένο αυτό θέμα θα επαναληφθεί η συζήτηση και στη συνάντηση, την επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Επίσης εγκρίναμε και το πρόγραμμά μας της επίσκεψης στην Ελλάδα από τις 27 μέχρι τις 29 Απριλίου. Σχετικά επίσης μιλήσαμε και την επιστολή προς τον κύριο Νταφ γύρω από τις εκτιμήσεις που έχουμε για το πώς πήγε δηλαδή η διαδικασία ακρόασης των επιτρόπων με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή στα σημεία που μας αφορούν. Για την επόμενη συνάντηση των συντονιστών θα πρέπει να μας δοθούν από όλες τις πολιτικές ομάδες οι μελέτες για το 2010. Κάποιες ομάδες το έχουν ήδη κάνει. Προβλέπεται επίσης να ορίσουμε και τους όρους ακροάσεων των νέων μελών του ελεγκτικού συνοδρίου, όπως επίσης και οι πρώτες συζητήσεις για τα προσχέδια προϋπολογισμού για το 2011. και επίσης ε, πρώτη ανταλλαγή επιστολών αποφασίστηκε γύρω από την ακρόαση στον τομέα της έρευνας μου έστειλαν ένα mail από τη γραμματεία, δεν ξέρω αν το πήρατε κι εσείς, λέγοντας ότι από τις 6 μέχρι τις 6.30 θα συνεχίσουμε την πρωινή συνεδρίαση, έτσι ώστε να πάρουμε κάποιες ε, αποφάσεις για τα θέματα στα οποία αναφέρθηκα ήδη. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε δηλαδή την τακτική μας συνεδρίαση την 18η απογευματινή. Θα ήθελα να χαιρετήσω λοιπόν τον πρόεδρο Καλτέρα για την παρουσία του και του δίνω αμέσως το λόγο για να παρουσιάσει το σημείο 19 της ημερήσιας διάταξης πρόγραμμα εργασίας για το 2010 του ελεγκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζει αγγλικά ο κύριος Πρόεδρος του συνεδρίου. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή μου που μπορώ να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2010. Το πρόγραμμα αυτό συνετάχθη από το ε, Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αισθάνεται τις διαρκείς επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης σε αυτή την περίοδο που βρίσκεται και πλήττεται η διακυβέρνηση, η οικονομική της διαχείριση. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών προσπαθούν να μειώσουν τις δαπάνες. Στόχος είναι να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα κονδύλια. Σε αυτή τη χρονική στιγμή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ανανεώνονται. Έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο, μια νέα συνθήκη και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτές ε, οι εξελίξεις θα συνεπιφέρουν έναν αριθμό ευκαιριών για να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ αυτών και η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, η αναθεώρηση του προπολογισμού και η προπαρασκευή για την περίοδο δημοσιονομικών προοπτικών από το 2014 και εφ' Το 2010 επίσης ανανέωση και για το ελεγκτικό συνέδριο, καθώς προσβλέπουμε στο να υιοθετηθούν νέοι κανόνες διαδικασίας μετά από την έγκριση εχθές από το Συμβούλιο, καθώς επίσης και το να καλωσορίσουμε νέα μέλη το 2010 το πρόγραμμα του ελεγκτικού συνεδρίου συμπεριλαμβάνει πολλούς στόχους που εμπλέκονται οι κυριότεροι δράστες για την εποπτεύση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και έχει προετοιμαστεί ευθυγραμμισμένα πάντα με τους στόχους της στρατηγικής για την περίοδο 2009-2012 που ε, είχε υποβληθεί και προς την κοινοβουλευτική σας επιτροπή πέρσι και εξακολουθεί να έχει τη σημασία της. Αυτή η στρατηγική στόχη του ελεγκτικού συνεδρίου στοχεύουν στο να μεγιστοποιήσουν τις επιπτώσεις ε, και να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων. Το πρόγραμμα εργασίας τονίζει τις προτεραιότητες του ελεγκτικού συνεδρίου. Περιγράφει τις εκθέσεις που θα δημοσιευθούν το 2010, καθώς επίσης και τις νέες εποπτικές και ελεγκτικές δραστηριότητες που θα ξεκινήσουν φέτος, που όμως στα επόμενα χρόνια θα αντανακλώνται σε εκθέσεις. Επίσης αναθεωρεί σε τακτά διαστήματα τις προτεραιότητες του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να γίνει η καλύτερη χρήση των πόρων. Όπως βλέπουμε στο πρόγραμμα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ταυτοποιήσει αρκετούς τομείς για την περίοδο 2009-2012 καθώς επίσης και συγκεκριμένες προτεραιότητες για το 2010 Μεταξύ αυτών είναι εκείνες που αφορούν την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τις κλιματικές αλλαγές, την αηφορία στην Ευρώπη, την Ευρώπη ως παγκόσμιο εταίρο και καλύτερες ε, διατάξεις, better regulation, καλύτερη νομοθεσία θα παρακολουθηθούν αυτά σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο των εκθέσεων και σε σχέση με τις την ετήσια έκθεση και τις ειδικέ εκθέσεις. Κύριε Πρόεδρε, ένα σημαντικό τμήμα των πόρων του κονδυλίου χρησιμοποιούνται για την δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης ε, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης. Αυτή η έκθεση συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα του έργου ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο, ιδιαίτερα την βεβαίωση αξιοπιστίας όσον αφορά την νομιμότητα όλων των συναλλαγών που εξετάζονται πέρυσι και φέτος το συζητούμε αυτό, στην ετήσια έκθεση του Συμβουλίου σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την γενική μείωση των αχρεωστήτων καταβληθέντων καθώς επίσης και όσον αφορά την, τον εντοπισμό θεμάτων που πρέπει ακόμα να ε, ε, ρυθμιστούν σωστά το έργο για το 2009 όσον αφορά τον έλεγχο βρίσκεται σε προηγμένη φάση και βρισκόμαστε σε ενεξελίξη διαδικασία. Στοχεύουμε στο να διευρύνουμε την έκθεση, την εποπτεία των πολιετών δαπανών, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάκτηση πληρωμών και τις ε, επανορθώσεις. Στην έκθεση του 2009 συνεχίζουμε να οικοδομούμε στην δομή που εισήχθη στην έκθεση του 2007. Αυτό το κεφάλαιο δίνει αξιόπιστα θεμέλια για συγκρίσεις μεταξύ ετών και μεταξύ τομέων πολιτικών. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζει το Ελεκτικό συνέδριο ότι υπάρχει χώρος και περιθώριο για βελτιωμένη απόδοση όσον αφορά την προσέγγισή μας και για την βελτίωση όσον αφορά την σαφήνεια και την συνεκτικότητα της ετήσιας έκθεσης. Προς αυτό το στόχο όπως είχα αναφέρει πέρυσι την ίδια χρονική στιγμή το Συμβούλιο με την υποστήριξη και εξωτερικών συμβούλων θα προσπαθήσει να, να εξετάσει τρόπους και οδούς με τους οποίους θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τους έλεγχους μας καθώς επίσης και τον επαναπροσδιορισμό της κάλυψης των συγκεκριμένων αξιολογήσεων. Έτσι το έργο θα υλοποιηθεί το 2010 ως προς αυτό το εγχείρημα. Επιπλέον το Συμβούλιο στοχεύει στο να δημοσιευθούν 40 ε, ειδικέ εκθέσεις ε, για τις ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οργανισμούς, κοινού οργανισμούς και άλλους φορείς. Ο αυξημένο αριθμός αυτών των φορέων και υπηρεσιών είναι μια αυξημένη πρόκληση όσον αφορά την επιπλέον εποπτεία που θα απαιτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθώντας να υλοποιήσει τους, τις υποχρεώσεις του, το ελεγκτικό συνέδριο έχει κονδύλια στον προϋπολογισμό του για να μπορέσει να ε, κάνει επιλεκτικούς ελέγχους και ε, ελέγχου συμμόρφωση που θα αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστών εκθέσεων. Επιλέγοντα αυτό το έργο λαμβάνει το Συμβούλιο ε, συγκεκριμένα στοιχεία υπόψη όπω του κινδύνου, το επίπεδο δαπανών που συνεμπλέκεται, την περίοδο που έχει ε, περάσει από προηγούμενου ελέγχου μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών αυτών προτεραιοτήτων προ όφελο του Δημοσίου. Όσον αφορά το πρόγραμμα 2010, συγκεκριμένε προτεραιότητε που εντοπίζονται από το Συμβούλιο είναι η πολιετής φύση των δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη και τις διορθώσεις και την ανάκτηση καινοτομία και εσωτερική αγορά, ανθρώπινο δυναμικό, αηφορία όσον αφορά τα ενεργειακά θέματα και απλουστευμένη στρατηγική για το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτού του, αυτού, του εγχειρήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνολικά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στοχεύει να δημοσιεύσει 20 ειδικέ εκθέσεις εφέτος Μέχρι το 2010 έχουν τυπωθεί τέσσερις τέτοιες εκθέσεις ε, όσον αφορά την κατάρτιση και εκπαίδευση των γυναικών, προενταξιακή βοήθεια στην Τουρκία, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, επίτευξη των στόχων των, οργαν... των υπηρεσιών του... Ε, των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και την επίτευξη των οικονομικών στόχων. Επίσης Εφέτος στοχεύουμε στο να δημοσιεύσουμε επιπλέον 16 εκθέσεις, εκείνες που ε, συσχετίζονται με τις κυριότερες προτεραιότητες, ε, την ανάκτηση υπό την κοινή αγροτική πολιτική, την ε, έρευνα και τις υποδομές, ε, μέτρα κινητό, μεγαλύτερης κινητικότητας και πρόγραμμα Λεωνάντο Νταβίντσι και το πρόγραμμα αξιολόγησης όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή επόπτευση της καλύτερης νομοθεσίας. Όσον αφορά το πρόγραμμα 2010, το Συμβούλιο στοχεύει να ξεκινήσει πέρα από αυτό ε, την εργασία σε στόχους για τους οποίους θα υπάρξουν εκθέσεις το 2011 ελέγχους ε, για θέματα όσον αφορά την διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου, μέτρα για να υπάρξει μείωση του υπερπλεονάζοντος δυναμικού στην, ε, στον αλλιευτικό στόλο. Κύριος στόχος όσον αφορά τις δραστηριότητες του Συμβουλίου για την περίοδο 2009-2011 είναι να αυξηθεί ο έγκαιρος χαρακτήρας και η ποιότητα όλων αυτών των ειδικών εκθέσεων που θα συντάσσονται. Το αναφέρω ως προς το εξής ο αριθμός των εκθέσεων ήδη αυξάνεται από 12 το 2008 σε 18 το 2009. Όμως αναγνωρίζει το Συμβούλιο ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για να βελτιωθεί η χρονική στιγμή υποβολής αυτών των εκθέσεων πιο έγκαιρα. Και με την αναθεώρηση των νέων κανόνων διεργασιών στοχεύουμε στο να υπάρξει ταχύτερη ε, διεργασία που θα διέπει την έγκριση και σύνταξη των ειδικών εκθέσεων. Επιπλέον και σύμφωνα με ευθυγράμμιση προς τις συστάσεις που έχουν υποβληθεί, το Συμβούλιο στοχεύει στο να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα των ελέγχων κατά το 2010 προβλέποντας την έναρξη σε ισχύ νέων διεθνών προδιαγραφών και ρητρών. Πέρα από τη σύνταξη εκθέσεων, το Συμβούλιο επίσης συντάσσει γνωμοδοτήσεις όσον αφορά τις ε, επιπτώσεις που ε, έχουν κάποια ε, μέτρα ή και αυτοβούλος συνεισφέροντας τον θεσμικό διάλογο και στα θέματα που βρίσκονται υπό συζήτηση δημόσια για τα δημόσια οικονομικά και το Συμβούλιο το 2009 έκανε μια αναθεώρηση της ετήσιας και των ειδικών εκθέσεων για να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι δηλαδή είναι οι κύριες προκλήσεις υπό το πρίσμα του ελεγκτικού συνεδρίου για να βελτιωθεί η οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή δημοσιεύθηκε ως γνωμοδότηση του Συμβουλίου μας υπαριθμών 1-2010 και θα υποβληθεί κατά λεπτό στη συνέχεια. Σημειώνω με ευχαρίστηση ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο στον πρόσφατο λόγο που εξεφώνησε προς την Ευρωβουλή ανέφερε κάποια από τα κυριότερα θέματα αυτής της γνωμοδότησης όταν είπε ότι η νέα Επιτροπή θα έπρεπε να επικεντρωθεί παράθεμα στην ποιότητα σε σχέση με τα κονδύλια και τις δαπάνες ώστε να υπάρχει πρόσθετη αξία και στο θέμα της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών και Εκείνο το οποίο ε, κατανοώ επίσης είναι το ότι αυτό το οποίο υπογραμμίστηκε χθε ε, στην Επιτροπή σας, η σημασία του να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την βελτιωμένη, την αναβάθμιση της ποιότητας ε, όσον αφορά τις δράσεις μας από πλευρά των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων. Το 2010 προβλέπουμε να υπάρξει γνωμοδότηση για τον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, καθώς περιορίζονται τα δημόσια κονδύλια διαθέσιμα, η βελτίωση της ποιότητας, η αναβάθμιση της ποιότητας του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτά τα κονδύλια αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Είναι περίοδος καινοτομία αυτή και καινοτόμων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα. Η συνθήκη ενισχύει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την το συνομοθετικό του έργο και έτσι το ελεγκτικό συνέδριο είναι το ανεξάρτητο ελεγκτικό και θεσμικό όργανο της Ένωσης. Γι' αυτό προσβλέπουμε εμείς ως Ελληνικό Συνέδριο στο να συνεργαστούμε στο μέλλον με την Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή υπό το πνεύμα αμοιβαίου σεβασμού, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα δραχθεί της ευκαιρίας η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και να βελτιώσει τα δημοσιονομικά της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν επιθυμεί κανεί ε, ευρωβουλευτή ή κυρία Γκρέσλε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την εντυπωσιακή επισκόπηση των όσων θα πρέπει να αναμένουμε στην επόμενη χρονιά. Και μάλιστα θα αυξήσετε τις εκθέσεις από 12 σε 20. Πολύ δουλειά επομένως για μας. Χαιρόμαστε. Βέβαια, αλλά πόσο. Πάντως εκτιμούμε πολύ το ότι επιθυμείτε να εργαστείτε σκληρά. Πάντως ε, επιθυμώ να σας ευχαριστήσω και εσάς και τα άλλα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου γιατί η προσπάθειά σας είναι αξιολογότατη. Όταν εκφράζω τέτοιες ευχαριστίες έχω να συνδέσω μια παράκληση. Χρειαζόμαστε συνεργασία γιατί τα προβλήματα μάλλον αυξάνονται παρά μειώνονται. Θα υπενθυμίσω ορισμένα θέματα όπου αντιμετωπίζουμε δυσχέρειες να λάβουμε πληροφορίες για την δήλωση αξιοπιστίας. Θα σας παρακαλέσω να εξετάσετε πώς μπορούμε να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα εκεί όπου προκύπτουν. Για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα, όπου δώσατε πράσινο φως τώρα. Αλλά στη Γερμανία έχουμε ένα περιθώριο σφάλματος 0,1 έως 0,3%. Σε άλλες χώρες είναι πάνω από 10%. Θα θέλαμε λοιπόν Αυτά τα έχουμε από τα νούμερα της Κομισιόν. Θα θέλαμε να έχουμε παρόμοια νούμερα, στοιχεία και από το ελεγκτικό συνέδριο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες. Γνωρίζω ποια είναι η κατάσταση όπως απορρέει από την συνθήκη και από το δίκαιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα στοιχεία, τα δεδομένα που διαθέτετε εσείς είναι ανεξάρτητα, για μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πόση σημασία έχουν τα ανεξάρτητα δεδομένα το γνωρίζουμε ιδίω από τώρα, από την περίπτωση της Ελλάδας και μετά. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν οι πληροφορίες που διαθέτεται σχετικά με την αξιοπιστία των στατιστικών δεδομένων που ανακοινώνουν οι χώρες μέλη να μας τεθούν υπόψη. Διότι απεδείχθη ότι οφείλουμε να είμαστε δύσπιστοι. Δεύτερη παράκληση. Οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας. Υπήρξε μέχρι τώρα πεδίο αγώνος εδώ για μας. Εσείς κάνατε μια σχετική ανακοίνωση, την οποία λάβαμε υπόψη. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να βασιστεί στα όσα διαθέτουμε και όπου να μπορούμε κάτι να κάνουμε και εμείς, δηλαδή να δράσουμε στη βάση του συστήματος αυτού, αλλά και οι χώρες μέλη. Δηλαδή να ενταχθούν οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας στους υφισταμένους ελέγχους. Όχι δηλαδή να μπει ακόμα ένα στρώμα ελέγχων, αλλά να γνωρίζουμε ότι αυτή στιγμή λάβουμε μια εθνική δήλωση αξιοπιστίας, μπορούμε πλέον να σταματήσουμε τους ελέγχους στο προκείμενο θέμα. Όχι να κάνουμε και άλλους ελέγχους. Χρειαζόμαστε λοιπόν την υποστήριξη του ελεγκτικού συνεδρίου για να δούμε πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα τέτοιο σύστημα. Μας είπατε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε εσά. Αυτό είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δεν είπατε όμως σχετικά με την συνεργασία με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Γνωρίζω ότι το θέμα αυτό είναι καυτό για σας. Αλλά εξηγήστε μας λίγο περισσότερο πώς εξελίσσεται η συνεργασία με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και πού μπορούμε εμείς να ε, λάβουμε κάποιες πληροφορίες, διότι εάν λάβουμε εν τέλει μια εθνική δήλωση αξιοπιστίας, αλλά αυτή δεν βασίζεται πουθενά, δεν βασίζεται σε δεδομένα δηλαδή των ελεγκτικών συνεδρίων, τότε δεν έχει απολύτως καμία αξία. Βεβαίως θα χρειαστεί να θεσπιστούν νέες διαδικασίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη, αυτό το γνωρίζω. Θα χρειαστούν λοιπόν στοιχεία καινοτομία. Αυτό πρέπει να γίνει όμως και για τι εθνικέ δηλώσει. Και μια παράκληση ακόμη. Επικρίνουμε από καιρού το σύστημα ανάκτηση. και αυτά που προτείνει το ελεγκτικό συνέδριο είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χθε είχαμε ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο της Περιφερειακής Ανάπτυξης Είχαμε παρακαλέσει το Ελεκτικό Συνέδριο να συνεργαστεί για να υπάρξει ένα ενιαίο σύστημα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα υπόψη μας. Το ερώτημα είναι πότε μπορούμε να αναμένουμε αυτά τα αξιόπιστα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης και για τα καλά σας λόγια. Είμαι ευγνώμων για την αναγνώριση αλλά και για την υποστήριξη. Επιτρέψτε μου τέσσερα σημεία να καταθέσω γύρω από τα σχόλια που κάνατε. Εμείς προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας ο στόχος του να δημοσιεύσουμε 40 εκθέσεις ειδικευμένε το 2010 θα δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες πρακτικά και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να το κάνουμε αυτό έτσι ώστε να είναι όσο περισσότερο εύχριστες γίνονται συνειδητοποιούμε ότι απαιτείται εν πάση περιπτώσει να κυκλοφορούν οι εκθέσεις αυτές σε έφετο χρόνο κάθε φορά και προσπαθούμε πάντα μέσω των εκθέσεων αυτών να σας δώσουμε την δυνατότητα να ξεπεράσετε τα προβλήματα και τους περιορισμούς του πιστοποιητικού αξιοπιστίας. Και έρχομαι εδώ στην πρώτη σας ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, θα πρέπει αυτά τα πιστοποιητικά να δίνουν την δυνατότητα να κατανοήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις χώρες, στις χώρες μέλη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Προσπαθούμε αυτά τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας να είναι πράγματι εύχριστα. Ο καλύτερος τρόπος όμως για να σας διαθέσουμε και στο Κοινοβούλιο να διαθέσουμε περισσότερες πληροφορίες ε, δεν μπορεί να είναι άλλος από τις εξειδικευμένες εκθέσεις, τα special reports του ελεγκτικού συνεδρίου για τα συστήματα χρηματοδότησης στη Γεωργία σαν παράδειγμα μέσα από τη δήλωση αξιοπιστίας δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη που έχετε για λεπτομέρειες, αλλά μέσα από την ειδική έκθεση για τη χρηματοδότηση στη Γεωργία μπορούμε. Τώρα για τα εθνικά συστήματα ελέγχου. Η συνεργασία μας με τα εθνικά συστήματα ελέγχου είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Δεν σας μεταφέρουμε εδώ κάτι το νέο, αλλά συνεχίζουμε να πιέζουμε στα πλαίσια της Επιτροπής Επαφής και Συνεργασίας για να καταλήξουμε σε μια κοινή αντιμετώπιση σχετικά με την δήλωση αξιοπιστίας. Ελπίζω να το πετύχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα σε όλους τους εθνικούς οργανισμούς που ασχολούνται με ελεγκτικές δραστηριότητες να δημοσιεύουν τις δραστηριότητες τους αυτές και τα προγράμματά τους χρησιμοποιώντας μια κοινή αντιμετώπιση. Και νομίζω ότι αυτό θα ξεκινήσει σε επίπεδο τακτικής και θα βοηθήσει το ελεγκτικό συνέδριο να καταλήγει στις σωστές αποφάσεις σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία του δίδουν τα εθνικά συστήματα ελέγχου. Προχωράμε ακόμα περισσότερο. Έχουμε συμφωνήσει να αναπτύξουμε διμερός συγκεκριμένες ελεγκτικές διαδικασίες, ιδιαίτερα στον τομέα γεωργίας, με τρία εθνικά ελεγκτικά συστήματα, έχοντας συμφωνήσει από πριν για τους τρόπους με τον οποίο θα κάνουμε την συγκεκριμένη επιτόπια έρευνα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι ακόμα πιο σημαντικό και από τη δήλωση αξιοπιστίας. Ο δρόμος είναι μακρύς και δεν μπορούμε παρά να σεβαστούμε τις εργασίες των εθνικών ελεγκτικών αρχών υπάρχουν ανησυχίε εκεί, υπάρχουν εθνικά ενδιαφέροντα, υπάρχουν συνταγματικοί περιορισμοί, είναι γενικά περίπλοκο τα θέματα. Γι' αυτό λοιπόν οι εθνικές δηλώσεις, και εδώ είναι σωστό να κάνουμε τη διάκριση από τις εθνικές δηλώσεις που υποβάλλουν ε, τα αρμόδια υπουργεία της κυβέρνησης, το Υπουργείο Οικονομικών σαν παράδειγμα, Εκεί είναι σαφές ότι το δικαστήριο θεωρεί, ότι μάλλον ε, το ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι οι δηλώσεις αυτές παρέχουν πληροφορίες και σχετικά με τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου τα οποία επικρατούν και χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες. Αυτού του τύπου οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας έχουν θετικά χαρακτηριστικά σε εθνικό επίπεδο όμως. Πρέπει να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο, να αναλυθούν σε εθνικό επίπεδο. Η τελευταία που διάβασα σαν παράδειγμα αφορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο, προήλθε μάλλον από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και έχει ελεγχθεί φυσικά η δήλωση αυτή από την αρμόδια υπηρεσία. και υπάρχει η δυνατότητα, προβλέπεται η δυνατότητα τα στοιχεία αυτά που θα δοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ίσως και κάποιες μορφές σε εισαγωγικά αποζημίωσης όταν διαπιστώνονται κάποια προβλήματα σοβαρά. Λοιπόν, οι εθνικές αυτές δηλώσεις έχουν κυρίως εθνικό στόχο χρήσης θα έλεγα. Παρόλα αυτά στα πλαίσια αυτής της εθνικής εικόνας αντίληψης ε, θα έλεγα για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα ίσως να δίνουν την δυνατότητα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τμήματα ε, των δηλώσεων αυτών. Τώρα, οι εθνικές δηλώσεις οι οποίες προέρχονται από τα εθνικά ελεγκτικά συστήματα και ιδρύματα σύμφωνα με προσυμφωνημένες μορφές εργασίας και συλλογής αρμοδιοτήτων. Τότε σε αυτή την περίπτωση το ελεγκτικό συνέδριο σαφώς και μπορεί να χρησιμοποιήσει με ευρύτερο τρόπο τις δηλώσεις αυτές. Υπάρχει και μία κατηγορία διαφορετική, μια τρίτη είναι οι λεγόμενες ετήσιες, ε, οι ετήσιες επισκοπήσεις των ελεγκτικών δραστηριοτήτων και χρησιμοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προορίζονται και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν ένα επιπλέον αν θέλετε συμπληρωματικό σύστημα δήλωσης αξιοπιστίας ένα επιπλέον στοιχείο που δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις ελεγκτικές διαδικασίες, να δει τι μαθήματα μπορεί να βγάλει από τις διαδικασίες αυτές, από τις αιτήσιες αυτές επισκοπήσεις. Οι επισκοπήσεις αυτές είναι ένα επιπλέον στοιχείο του εθνικού ελεγκτικού συστήματος και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αυτά και αφορούν κυρίως φυσικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι κάτι το οποίο το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσει εκ των υστέρων. Όπως είπα και νομίζω ότι είναι σωστό αυτό, δεν θα πρέπει να δημιουργούμε επικαλύψεις συνεχής στα πλαίσια των ελεγκτικών συστημάτων. Και ήδη έχουμε να αντιμετωπίσουμε υπερελεγκτικές καταστάσεις θα έλεγα σε ορισμένους τομείς και αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ε, να χρησιμοποιούμε σωστά τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χρησιμοποιώντας όλη την προστιθέμενη αξία που μας δίδουν οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας όλων των ειδών όπως είπα. Τέταρτο στοιχείο είναι το στοιχείο ανάκτησης και εδώ τίθεται το θέμα της αξιοπιστίας της πληροφορίας, της αξιοπιστίας των στοιχείων τα οποία μας δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήθως. Εμείς εδώ πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση όσο επιφυλακτικοί και ανήμεθα να αντικαταστήσουμε την υπευθυνότητα και να αναλάβουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει και στα πλαίσια της ε, εφαρμογής της νέας συνθήκης να δούμε πώς ε, θα γίνουν οι αλλαγές στο δημοσιονομικό κανονισμό σύμφωνα με τη νέα συνθήκη. Υπάρχει μια απόχρωση γιατί λέγεται ότι ασκείται ο προϋπολογισμός, εφαρμόζεται ο προϋπολογισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα άλλα όργανα. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει κάτι τέτοιο. Θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη σαν παράδειγμα να υπάρξουν περισσότερες καταστάσεις, δηλαδή ουσιαστικά θα εμβήσουμε συνταγματικά την ισχύουσα κατάσταση σχετικά με τον σημαντικό ρόλο που έτσι και αλλιώς παίζουν τα κράτη-μέλη. Πώς αυτό θα περάσει, πώς θα εφαρμοστεί στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό μένει να γίνει. Και ακριβώς και μέσα από τη Νέα Συνθήκη αυτά τα οποία έχουμε πει για τις ετήσιες επισκοπήσεις και τις δηλώσεις αξιοπιστίας νομίζω ότι όλα αυτά τα μέσα δεν μπορούν παρά να βοηθήσουν να λειτουργήσουμε καλύτερο. Κύριος Ριμπεράτσκι. Ο πρόεδρος κύριος Καλντέρα είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και τον άκουσα με πάρα πολύ προσοχή. Άκουσα λοιπόν και συγκεκριμένα τα στοιχεία που ανέφερε για το πρόγραμμα του οργάνου του για το 2010. Να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις, ίσως χρήσιμες για τη συζήτηση και στα πλαίσια της διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής για το έτος 2008. Πριν από οτιδήποτε άλλο θα ήθελα να χαιρετήσω το ξεκαθάρισμα των προτεραιοτήτων για το 2010. Είναι πέντε οι προτεραιότητες αυτές, είναι πραγματικές προτεραιότητες, δεν είναι ένας τεράστιος κατάλογος χωρίς τέλος, γιατί όταν είναι πολλές οι προτεραιότητες πάβουν ουσιαστικά να είναι τέτοιες. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα το κεφάλαιο το οποίο αναφέρατε, το οποίο ονομάζεται νέα προϊόντα, new products είναι αλήθεια ότι έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια νέα πρόταση από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου για νέες μορφές εργασίας. Και εδώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα κύριε Πρόεδρο. Συζητήσαμε το θέμα της απαλλαγής για το 2008 και ασκήθηκαν κριτικές από πλευρά των μελών της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου για την δειγματοληψία, το λεγόμενο sampling. Εμείς δεν αμφισβητούμε την μέθοδο αυτή, την μέθοδο εργασίας, αλλά για να απλουστεύσουμε λίγο τα πράγματα, καλό θα ήταν να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί για μας, νομίζω, έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουμε τα επιχειρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μέθοδο της δειγματοληψίας. Δεν εκφράζουμε επιφυλάξεις σχετικά με τη μεθοδολογία. Ε, συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι τέλεια η μεθοδολογία αυτή. Αλλά εφόσον χρησιμοποιηθεί με τακτό τρόπο σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, σαφώς και μας επιτρέπει να διακρίνουμε την πορεία των τάσεων. Αναφερθήκατε επίσης και στην έκθεση σε κίνδυνο και τους κινδύνους που υπάρχουν. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το περιθώριο κινδύνου στο οποίο αναφέρεται η Επιτροπή. Υπάρχει ένα τέτοιο περιθώριο κινδύνου. Σαν παράδειγμα, το περιθώριο αυτό για το Ταμείο Συνοχής είναι διαφορετικό από ότι για τα διαρθρωτικά ταμεία. Φαίνεται ότι για το Ταμείο Συνοχής σαν παράδειγμα δεν είναι τόσο υψηλό. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο κινδύνου. Ο κίνδυνος αυτός μερικές φορές μπορεί να είναι αποδεκτός, μερικές φορές μπορεί να είναι αναμενόμενος, μερικές φορές μπορεί να χαρακτηρίζεται σαν ανεκτός, το επίπεδό του να χαρακτηρίζεται σαν ανεκτό περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ήθελα επίσης περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα λεγόμενα πολιετή, με τις πολιετής δαπάνες, δηλαδή επαναλαμβανόμενες ετήσια βάση δαπάνες. Τι συνεννόηση υπάρχει γύρω από αυτό με τα κράτη-μέλη. Τι σχέση έχουν αυτές οι δαπάνες και πώς συνδέονται με τις κοινοτικές δραστηριότητες. Μπορούμε να έχουμε διαίρεση σε επίπεδο ποσοστώσεων των δαπανών αυτών. Ιδιαίτερα όταν βλέπει κανείς τον τρόπο που κατανέμονται τα διαφθορτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, μερικές φορές δεν ξέρουμε. Υπάρχει μια σύγχυση από την πολυδιάσπαση, υπάρχει μια διαδοχική σώρευση των χρήσεων των συγκεκριμένων πιστώσεων και υπάρχει μια έντονη σύγχυση. Δεν ξέρουμε για το τελικό ύψος του ποσού για το οποίο μιλάμε. Είναι 7 ε, εκατομμύρια, 14 εκατομμύρια ανά περίπτωση. Για την κυρία Γκρέσλα, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε, διαφθρωτικά ταμεία, όπως επίσης και ταμείο συνοχής, όπως επίσης και μέθοδοι ανάκτησης. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση για τις εξελίξεις και τις τάσεις των ταμείων αυτών. Ήδη προσπαθούμε να διατυπώσουμε μια πρόταση στο όνομα του Προέδρου μας, μια έκθεση ουσιαστικά, Θέλουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για την παρουσία σας. Ελπίζω να απαντήσετε σε αυτά που ρώτησα. Λοιπόν, θα ακούσω και άλλους αν έχουν κάποιες ερωτήσεις και θα κλείσει μετά ο πρόεδρος του ελεγκτικού. Η κυρία Ολμαγερ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σας ευχαριστώ πρώτα-πρώτα για την παρουσία σας εδώ. Είμαι νέα Ευρωβουλευτής και χαίρομαι για το γεγονός ότι το ελεγκτικό συνέδριο υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε τέτοιο βαθμό. Βρίσκω ενδιαφέρουσα την έκθεσή σας και για τις εκθέσεις που προτίθεστε να κάνετε θα ήθελα να συνδέσω μια παράκληση. Εμφανίστηκε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα και προσεκτικά. Στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές το έχουν διαπιστώσει και άλλοι συναδελφοί μου άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων και αναφέρομαι στο πρόγραμμα ΣΥΣ 2 ένα πρόγραμμα που έχει σχέση με την συμφωνία του Σέγγεν και το οποίο βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού εδώ και μία οκταετία. Και τώρα πάλι μετά από μια πρώτη αφετηρία κατέρευσε το σύστημα μετά από 26 ώρες με δαπάνη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και με μηδενισμό της μέχρι τώρα μεγάλης και βαριάς εργασίας που έχει καταβληθεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι λαμβάνει εν λευκό επιταγές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω διαδικασία και το προγραμματισμό του ΣΥΣ 2. Αυτό όμως δεν ικανοποιεί τους ευρωβουλευτές. Για πολλούς και πολλέ από τους συναδέλφους μου διαφόρων πολιτικών κομμάτων και από τις συζητήσει που έχω κάνει μαζί τους προκύπτουν οι επιθυμίε τους να ελέγξει το ελεγκτικό συνέδριο πώς ήταν δυνατόν να προκύψει αυτό να εξεταστεί εάν έχουν υπάρξει ανομαλίες στις προσκλήσει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και άλλες δημόσιες προκηρύξεις και όπως είπα βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασίας εδώ και 8 χρόνια. Υποσχέθηκα στις και στους συναδέλφους μου ότι θα σας θέσω υπόψη την παράκληση αυτή σήμερα διότι πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα το οποίο έχει απόλυτη ανάγκη να διαλευκανθεί ώστε να μπορέσει και η δική μας Επιτροπή να σχεδιάσει για το μέλλον τις επόμενες ενεργές της. Σας ζητώ συγγνώμη που τώρα έρχομαι σε τόσο σύντομη προθεσμία και σας φορτώνω ακόμα ένα θέμα ενώ έχετε ήδη ετοιμάσει τον σχεδιασμό σας για τον επόμενο χρόνο. Μόλις προ δύο ωρών προέκυψε το θέμα αυτό από την συζήτηση που είχαμε τους άλλους συναδέλφους μου και γι' αυτό βεβαίως σας το θέτω υπόψη σας έτσι απότομα. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, δίνω το λόγο στον Πρόεδρο. Ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ολμάιερ γιατί και εγώ το ίδιο ήθελα να θέσω υπόψη σας, βέβαια ίδια το έθεσε με πολύ πιο γοητευτικό τρόπο, πάντως πρόκειται για μια κατάσταση όπου αφενός την αντιμετωπίσαμε πολύ βραχυπρόθεσμα, τέθη υπόψη μας δηλαδή, από την άλλη μεριά δεν είναι και η πρώτη φορά όπου από τις τάξεις των διαφόρων προσώπων που ασχολούνται στην πράξη με τα θέματα αυτά μου τονίζετε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις τράπεζες δεδομένων, με τα μηχανογραφικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου, πώς να το πω, να το πω έτσι διπλωματικά, έχουν ατυχήσει. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε απαιτεί διαλεύκανση. Κατά τη γνώμη μου το καταλληλότερο όργανο για να κάνει τη διαλεύκανση αυτή είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε τα πράγματα αυτά. Και στο πρόσωπό μας θα βρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικούς συμμάχους. Ασφαλώς τηρώντας απολύτως τις διατάξεις που εξασφαλίζουν την κυριαρχία του ελεγκτικού συνεδρίου. Παρ' όλα αυτά, διαρωτώ με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί μια συνέργεια των οργάνων μας για την διαλεύκανση τέτοιων καταστάσεων και να βελτιωθεί μάλιστα αυτή η συνέργεια στο μέλλον. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στο ελεγκτικό συνέδριο που τίνει πάντοτε ευήκον ους στις αιτήσει της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού και εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας θα σας πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και από την προθυμία που έδειξαν πάντοτε τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου να απαντούν στις ερωτήσεις μας στην Επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμού, αλλά και να είναι στη διάθεσή μας και για ανεπίσημες συζητήσεις, όπου μπορούμε ίσως να πούμε περισσότερα πράγματα και να δούμε πώς είναι δυνατόν ίσως να προταθούν κάποιες βελτιώσεις από πλευράς Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό διευκολύνει το έργο μας, νομίζω πάρα πολύ Ήρθα με κάποια καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη για την καθυστερημένη έλευσή μου, αλλά οφείλονταν στο ότι έκανα μια διάλεξη σε 50 νεαρές και νεαρούς δημοσιογράφους, όπου είπα ότι τα βέλη που έχουμε στο πλωστάσιο μας, στη φαρέτρα μας εμείς της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, μας τα έχει βάλει το ελεγκτικό συνέδριο και γι' αυτό λέω ότι η συνεργασία μαζί σας είναι τόσο πολύτιμη. Έχω μια ας πούμε μετριοπαθή πρόταση, η οποία έχει το εξή νόημα. Σχετικά με το χρονικό σημείο όπου υποβάλλεται η ετήσια έκθεση, το φθινόπωρο, γύρω στο Νοέμβριο δηλαδή, αν μπορούμε να εγγράψουμε στην ημερήσια διάταξή μας ένα θέμα όπου να επαναεπισκοπήσουμε, αν θέλετε, τους τελευταίους 12 μήνες και να υποβάλουμε, να θέσουμε υπόψη δηλαδή του ελεγκτικού συνεδρίου θέματα που για μας είναι καυτά. Θα ήθελα να μάθω κύριε Πρόεδρε, εάν θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο και αν αυτό θα σημάνει κάποια ενδιαφέρουσα για σας εισρωή, input θεμάτων από πλευράς μας για την ετήσια έκθεσή σας. Κύριε Αντρέας, ευχαριστώ κύριε Καλδείρα για την παρουσίασή σας. Για πάρα πολλά χρόνια το επίπεδο παρατυπιών στις πληρωμές και στις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσής δικαιολογεί λόγω της περιπλοκότητας των κανόνων ελέγχου. Δεν έγιναν όλα αυτά τα χρόνια πολλά πράγματα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Το ερώτημα είναι λοιπόν, μέσω της προσπάθειάς σας, έχετε συνειδητοποιήσει τα παραδείγματα και τους τομείς τους οποίους θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή των κανόνων. Μήπως θα πρέπει να δημοσιεύσετε ένα μνημόνιο με τις περιπτώσεις τις οποίες έχετε παρέμβει για να διορθώσετε τις παρατυπίες έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους να μας απαλλάξει από τα προβλήματα αυτά που τρέχουν χρόνια τώρα. Κύριε Καλντέιρα, κλείνετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλες σας τις ερωτήσεις. Θα είμαι συντομότερος από ό,τι πριν. Για τις ερωτήσεις του κυρίου Λιμπεράτσκι Θα επιμείνω σε ένα θέμα που θεωρώ κρίσιμο. Το ελεγκτικό συνέδριο χρησιμοποιεί μία θα έλεγα σαφέστατη μεθοδολογία που βασίζεται στα διεθνή επίπεδα τα ελεγκτικά. Ακολουθούμε αυτά τα διεθνή επίπεδα ελέγχου. Και η μεθοδολογία την οποία ακολουθούμε περιλαμβάνει επίσης και τη δειγματοληψία και όλα τα άλλα τα στοιχεία τα οποία επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε από τη δήλωση αξιοπιστίας. Προφανώς και αλλάζουμε και ανανεώνουμε τη μεθοδολογία μας. Παρ' όλα αυτά εμείς λειτουργούμε ελεγκτικά και χρησιμοποιούμε ακριβώς τα διεθνή ελεγκτικά στάνταρτς για να το κάνουμε. Λαμβάνω υπόψη τις ανησυχίες που υπάρχουν για την βοήθεια που θα πρέπει να δοθεί προς ε, το ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων τα οποία χρησιμοποιεί. Αλλά επαναλαμβάνω, αλλά ότι μάλλον τα δεδομένα τα οποία παρέχουμε και οι πληροφορίες τις οποίες εμείς παρέχουμε δεν είμαστε εμείς που τα συλλέγουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μας δίδουν τα στοιχεία αυτά. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάθε αίτημα του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σας για συγκεκριμένες εκθέσεις και για συγκεκριμένα θέματα. Αυτό δεν θα συμβεί για πρώτη φορά και ούτε και για τελευταία. Έχει μεγάλη σημασία όμως τα αιτήματα αυτά να τεθούν γραπτά, συγκεκριμένα δηλαδή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σύμφωνα πάντα με τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές μας να σας ικανοποιήσουμε. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για την ετήσια συνάντηση της Επιτροπής σας και των μελών τη συνάντηση ανάμεσα σε εσά και τα μέλη δηλαδή του ελεκτικού συνεδρίου. Το κάναμε αν θυμίστε και το Σεπτέμβριο του 2009 και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή έτσι ώστε να προσπαθήσουμε εμείς να κατανοήσουμε καλά στο ελεγκτικό συνέδριο της δικής σας ανησυχίες, τι απαιτήσει έχετε στα πλαίσια της προετοιμασίας του προγράμματός μας να προσπαθήσουμε να τις λάβουμε υπόψη μας, και πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε σαν παράδειγμα έχουν προταθεί από μέλη της Επιτροπής σας ή από τον προηγούμενο πρόεδρό σας. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι αποδεικνύουμε ότι είμαστε απόλυτα δεκτικοί στις ανάγκες σας και στις προτάσεις σας, στον βαθμό βέβαια των δυνατοτήτων μας και στον βαθμό των δυνατοτήτων του δυναμικού μας, σε βάση περιπτώσει, ε, το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Μία τελευταία πληροφορία. Να συνδυάσω δύο ερωτήσεις, μία της κυρίας Ανδρέασεν και του κυρίου Λιμπεράτσκι. Είπαν τι κινδύνους μπορεί να ανεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι μπορεί να βοηθήσει, πώς μπορεί να βοηθήσει το συνέδριο, το ελεγκτικό και το συνέδριο, λέει η κυρία Ανδρέασεν, θα πρέπει να πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρέπει να αλλάξει και πού. Εμείς δίνουμε παραδείγματα των προβλημάτων τα οποία διαπιστώνουμε σαν ελεγκτικό συνέδριο και προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Στον παράδειγμα, ο τομέα της έρευνας. Οι νέοι κανόνες για το 7ο πρόγραμμα έρευνας. Οι κανόνες αυτοί εν πολλής έχουν εμπνευστεί από τις προτάσεις οι οποίες συστηματικά γίνονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Αντιδρούμε επίσης αν οι προτάσεις τις οποίες κάνουμε αγνοούνται. Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως και το Κοινοβούλιο κατά τομέα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή συστημένων αλλαγών. Και εσείς σαν Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο είσαστε υπεύθυνοι και για την ομοθετική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά εμείς σας προτείνουμε τις βέλτιστες δυνατές μεθόδους και εσείς αποφασίζετε σε επίπεδο κοινοβουλίου, επιτροπής και συμβουλίου, ακόμα δε και κρατών μελών θα έλεγα. Η νέα συνθήκη δίνει σας θυμίζω στα εθνικά κοινοβούλια νέες αρμοδιότητες σχετικά με τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα σας δίνουμε στοιχεία, θα σας δίνουμε παραδείγματα, το έχουμε ήδη κάνει μέχρι τώρα, αλλά το ελεγκτικό συνέδριο από μόνο του δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Η μοναδική αρμοδιότητα την οποία έχουμε, η μοναδική να το πω αλλιώ εξουσία την οποία έχουμε είναι η της συστάσεως εξουσία. Και αυτό κάνουμε. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και τα πράγματα λοιπόν για το πώς θα πάνε εξαρτάται και από τα άλλα όργανα. Σωστή συνεργασία λοιπόν διοργανική είναι προαπαιτούμενο, είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο και να βελτιώσουμε την οικονομική διαχείριση στο εσωτερικό της Ένωσης. Ευχαριστώ τον πρόεδρο κύριο Καλντέιρα για την παρουσίαση του προγράμματος 2010 και για τις απαντήσεις τις οποίες έδινε. Περνάμε στο σημείο 20. Γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου σε σχέση με τη βελτίωση ε, της δημοσιονομικής διαχείρισης. Ο αρμόδιος επίτροπος, κύριος Μπονιτσί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι εδώ ανάμεσά σας και ανταλλάσσουμε κάποιες πρώτες απόψεις. Θα πρέπει να πω ότι όπως είπε και ο, προηγούμενος, ο πρόεδρος μας προηγουμένως, η λογική που οδήγησε στο έγγραφο αυτό, ή μάλλον να το πω αλλιώς η γέννηση του εγγράφου αυτού προκλήθηκε ουσιαστικά από σας από δικό σας αίτημα, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις που έχουμε στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαχείρισης. Μιλάμε για ένα μικρό κείμενο, 7-8 σελίδες. Προσπαθούμε να είμαστε συνθετικοί και συνοπτικοί και ελπίζουμε μέσα από το έγγραφο αυτό η Επιτροπή θα το διαβάσει προσεκτικά και εσείς προσεκτικά θα το διαβάσετε είμαι βέβαιος, δεν θα περιοριστείτε σε μια μικρή περίληψη από πλευράς των βοηθών σας, γιατί επιμένουμε σε κάποιους τομείς οι οποίοι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το μέλλον. Η Επιτροπή ήδη από το 1999 ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα διοικητικών αλλαγών για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης. Mm. Έχουμε τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας σήμερα, τις οποίες δεν είχαμε κάποτε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο το ελεγκτικό συνεδρίο έχει πράγματι σημειώσει βελτιώσεις στα πλαίσια του δημοσιονομικού ελέγχου και υπάρχει και μία σημαντική μείωση, μία διακριτή μάλλον μείωση των παρατυπιών. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν υψηλά επίπεδα λαθών σε ουσιαστικούς τομείς του προϋπολογισμού. έχουν, ε, τα στοιχεία είναι γνωστά της ετήσιας έκθεσης και μετά από τις συζητήσεις τις οποίες κάνατε και χθε, νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθω λίγο για ένα μικρό χρονικό διάστημα γιατί ίσως να δημιουργήθηκαν κάποιες απορίες. Αν δει κανεί την πρώτη στήλη, η πρώτη στήλη αφορά την αξιολόγηση των ελεγκτικών συστημάτων. Αυτά είναι δηλαδή τα βασικά στοιχεία τα οποία δείχνουν αν τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούμε λειτουργούν σωστά. Εκτός από δύο τομείς, στα έσοδα από τη μία και τις διοικητικές δαπάνες που δεν ξεπερνούν το 6%, το υπόλοιπο των δαπανών την χάνει μίας επιμέρους αποτελεσματικής ταξινόμησης. τα συστήματα κατελάχιστον τα οποία χρησιμοποιούμε, τα συστήματα που είναι διαθέσιμα σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οφείλουν να είναι αποτελεσματικά. Όταν λέμε ότι είναι επιμέρους αποτελεσματικά, αυτό σημαίνει ότι οι ελεγκτικές διαδικασίες δεικνύουν ότι υπάρχουν προβλήματα σε ορισμένους τομείς. Υπάρχει πολλή δουλειά λοιπόν η οποία μένει να γίνει και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι κι αλλιώς ένα μεγάλο ποσοστό των πιστώσεων είναι αντικείμενο κοινή διαχείρισης και από την Επιτροπή και από άλλα όργανα. Και το θέμα είναι να ελέγχεται η πληρωμή των πιστώσεων στον τελικό χρήστη, σε αυτόν, ο οποίος, ε, σε αυτόν για τον οποίο προορίζονται τα χρήματα. Και εδώ οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν είναι πολλές και απαιτούνται κοινέ δράσεις. Δεν ξέρω πόσο κοστίζουν αυτά τα συστήματα ελέγχου. Πάντως θα έχουν ένα συγκεκριμένο σοβαρό κόστος νομίζω. Υπάρχει ε, η λογική της, ε, του έλογου κόστους. Είναι πραγματικά η σχέση κόστους-οφέλους συμφέρουσα σε αυτή τη φάση. Ίσως όχι. Οι ετήσιες εκθέσεις, οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας μας δίνουν κάποια επιμέρους στοιχεία αλλά ίσως θα πρέπει να είμαστε λίγο περισσότεροι επιφυλακτικοί και ίσως αυτές οι πληροφορίες να είναι λίγο υπεραισιόδοξες. Σαν παράδειγμα στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης είχαν τεθεί κάποια προβλήματα σχετικά με δαπάνες στην Ελλάδα και είχαν υπάρξει επιφυλάξεις σε κάποιες από αυτές τις δαπάνες οι οποίες ήρθησαν εκ των υστέρων από πλευρά της Επιτροπής. Εμείς θέτουμε το ερώτημα. Υπήρξαν αρκετά στοιχεία τα οποία να επιτρέπουν την άρση των επιφυλάξεων. Ίσως να πιστεύουμε ότι εμείς δεν, ε, από τα στοιχεία τα επιπλέον που έχουμε δεν αποδεικνύεται ότι είναι επαρκή έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η άρση των επιφυλάξεων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα και στην, επιστολή σας, στην αποστολή σας συγγνώμη, στην Ελλάδα σαν παράδειγμα τέτοιου είδους ε, ε, θέματα θα τα αντιμετωπίσετε. Τα συστήματα αυτά είναι συστήματα λειτουργικά και έχουμε κάποιο περιθώριο λάθος αλλά δεν μπορούμε να κολλήσουμε στα πλαίσια αυτού του περιθωρίου λάθος πρέπει να το ξεπεράσουμε και να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα συγκεκριμένα προβλήματα. Στη δεύτερη στήλη, βελτιώσεις σημειώνονται στη Γεωργία, ειδικά στη Γεωργία. Υπάρχουν επιπλέον προκλήσεις βέβαια. Υπάρχουν κάποια νέα κρατημέλη τα, για τα οποία έχουμε περιορισμένα στοιχεία και ίσως θα πρέπει να δούμε καλύτερα τα συστήματα τα οποία υπάρχουν στις χώρες αυτές έτσι ώστε το ελάχιστο ποσοστό θα έλεγα λαθών και παρατυπιών να διαπιστώνεται. Υπάρχει μια μικρή μείωση επίσης των προβλημάτων και στη συνοχή. Αν δείτε σε επιμέρους κεφάλαια φτάνουμε στο 11%. Ανησυχώ εδώ λιγάκι. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι ένα τουλάχιστον 11% σε στατιστικό επίπεδο. Τι εννοούμε δηλαδή. Είμαστε δηλαδή κατά 95% ε, πεπισμένοι, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, ότι τουλάχιστον το 11% των πληρωμών δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει. Επί τη βάση των στοιχείων τα οποία είχαμε. Όλα αυτά βέβαια αφορούν την παλαιά προγραμματική περίοδο του 2000 με 2006 και ε, παρόλα αυτά τουλάχιστον το δύο, τα δύο τρίτα των δαπανών τις οποίες εξετάζουμε αναφέρονται σε αυτή την περίοδο την εξαετή, την παλαιά. Και μέσω των λεγόμενων μήνυντας νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί προσπάθησε να βελτιώσει κάπως τα πράγματα εσωτερικά, προσπάθησε να αναλάβει ένα επιπλέον ελεγκτικό ρόλο χωρίς να είναι όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο πραγματικός ελεγκτής και τα στοιχεία αυτά που χρησιμοποιούμε φτάνουν μέχρι τον μήνα Μάιο του 2009. Εν πάση περιπτώσει, περιορισμοί υπάρχουν σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα των στοιχείων και πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, παρά τις διαφορές σε σχέση με την προγραμματική περίοδο, βλέπουμε ότι έχουν υπάρξει με λίγα λόγια βήματα προόδου. Δεν μπορούμε να περάσουμε σε ποσοτική αξιολόγηση και εκτίμηση αυτών των βημάτων προόδου. Νομίζω ότι οι προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, ε, ε, πρέπει να επενεθούν, αφορούν όμως ίσως κάποιους τομείς δεν αναφέρονται σε θέματα τα οποία καλύπτονται σαν παράδειγμα και καθίστανται περιπλοκότερα μέσω του financial engineering κάποιων ρυθμίσεων χρηματοπιστωτικών. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κοιμηθούμε ήσυχοι μόνο και μόνο βλέποντας κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί πάντα. Και γι' αυτό καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναλάβει τις προσπάθειες που έκανε και τον επόμενο χρόνο. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και χρησιμοποιώντας περισσότερο βάθος σε επίπεδο λεπτομέρειας και αυτό θα βοηθήσει πολύ την κατάρτιση των εκθέσεων ετησία δραστηριότητας. Όταν υπάρχουν προβλήματα στον ελεγκτικό τομέα, αυτό το οποίο πάρα πολύ συχνά γίνεται είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε focus testing, δηλαδή συγκεκριμένη έλεγχη σε συγκεκριμένους τομείς. Σε συγκεκριμένους τομείς, σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένα προγράμματα, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά αυτό το focus testing στην ουσία έχει σαν στόχο την ανείχνευση των νέων προβλημάτων. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα και θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα σαν μέθοδο και οι γενικοί διευθυντές στην Επιτροπή. Ελεκτικές δραστηριότητες γίνονται. Ελεκτικές δραστηριότητες συμβαίνουν πάντα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Ιδιαίτερα στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περίοδου και ιδιαίτερα στα διαφορετικά ταμεία. Χρήσιμο θα είναι λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα και εδώ αυτό αφορά και τις ερωτήσεις αυτό το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν. Θα θέλαμε το ελεγκτικό συνέδριο να μας διαθέτει περισσότερες πληροφορίες. Είτε ένα κράτος μέλος είναι δύσκολο αυτό να γίνεται βέβαια λόγω των περιορισμένων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα έλεγα όμως αυτό είναι ένα σημαντικό εγχείρημα για τη διαχείριση, για την διακυβέρνηση. Να είναι κανείς σε θέση να λάβει καλύτερα υπόψη και να δει το τι συμβαίνει με αυτά τα κονδύλια σε σχέση με συγκεκριμένες χώρες ή συγκεκριμένα προγράμματα και για αυτούς τους λόγους να δούμε ποια διορθωτική, επανορθωτική δράση θα απαιτεί το να ληφθεί. Τώρα, το με υψηλό ποσοστό παρατυπιών, όπως είδατε, συνοχή, εξωτερική βοήθεια, ανάπτυξη, διεύρυνση και ίσως σε μικρότερο βαθμό ο τομέας της έρευνας και η νέα προγραμματική περίοδος καταδεικνύει κάποιες βελτιώσεις και το ανέφερε ο κύριος Καλντέρα πιο πριν και μας εκπλήσει κάπως ότι μέσω της, η ανάπτυξη της υπαίθρου δείχνει βελτιώσεις. Καλό αυτό. Όμως βρίσκονται πάλι σε υψηλό επίπεδο αυτά τα ποσοστά προσπαθήσαμε σε κάποιες λίγες γραμμές να εντοπίσουμε ποιες είναι οι περισσότερες ατυπίες, παρατυπίες που είδαμε. Για παράδειγμα, μη, αχρεωστήτως καταβληθέντα, μη συμμόρφωση, για παράδειγμα, με όρους για καταβολή πληρωμών, προβλήματα με τις δημόσιες προμήθειες, και αγορές. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας μείζον τομέας που ίσως θα έπρεπε να απλουστευτεί περισσότερο. Όλες οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη θα έλεγα έχουν κανονισμούς και διατάξεις για τις δημόσιες προμήθειες και μεγάλο μέρος των κονδυλίων του προϋπολογισμού περνά μέσω αυτών. Γιατί να είναι πρόβλημα λοιπόν να, μπορέσουμε, να μην μπορέσουμε να δούμε το τι γίνεται με τους κοινού ε, κανονισμούς και διατάξεις όσον αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειες. Πρέπει να το δούμε. Είναι ένα πρόβλημα. Αν δούμε τον τομέα των διαθωτικών ταμείων, αυτός είναι ένας τομέας που έχει προκαλέσει προβλήματα και οι δύο κυριότεροι, θα έλεγα, συντελεστές προβλημάτων σε σχέση με τον έλεγχο των κινδύνων και τον καθορισμό των αποδεκτών αυτής της βοήθειας, όπως αναφέρεται στην πρώτη ε, στήλη, και το θέμα των κανονισμών και διατάξεων επιλεξιμότητας. Και πράγματι, οι συνάδελφοι, είναι περίπλοκοι, σύνθετοι αυτοί οι κανόνες. Είχαμε τον Ισπανό Υπουργό εχθές που είπε ότι δεν μπορούμε να πλουστεύσουμε υπερβολικά αν δεν θέλουμε να χάσουμε, να απολέσουμε κάποια στοιχεία κατεύθυνσης ε, των κονδυλίων των ταμείων σε επιτέλεση συγκεκριμένου έργου. Καμιά φορά όμως διαρωτώμε αν έχουμε περίπλοκους κανόνες, αν μπορούν με το σωστό τρόπο να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αν έχουμε τόσο περίπλοκους και σύνθετους κανονισμούς. Αυτό είναι το δίλημα, το πρόβλημα το οποίο τίθεται και νομίζω υπάρχει αρκετό εύρος, αρκετό περιθώριο να σημειωθούν βελτιώσεις. Πώς να μειωθούν οι παρατυπίες. Όπως είπα στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, όπως αναφέρθηκε εκεί, πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Είναι μια εξαιρετική ε, εξέλιξη αυτή, προς τη σωστή κατεύθυνση εξέλιξη το ότι οι γενικοί διευθυντές πρέπει να υποβάλουν αυτές τις εκθέσεις δραστηριοτήτων για να δούμε κατά πόσο βαίνουν καλά τα πράγματα. Όμως υπάρχει μη επαρκής αξιολόγηση ίσως του προβλήματος καμιά φορά. υπερβολικά αισιόδοξα στοιχεία, οι συντελεστές που παρισφρέουν. Και όπως ανέφερα στην περίπτωση της Ελλάδας για παράδειγμα, για το, προτού τα αποτελέσματα τα έχουν, να έχουν ε, διαβιβαστεί ήρθε ο περιορισμός και αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο ικανοπτικό τώρα βελτίωση των μηχανισμών για τις ανακτήσεις όσον αφορά το στοιχείο αυτό ακούσατε χθε ε, κάποιες εκτιμήσεις για τις ανακτήσεις η μόνη έλεγχη για αυτά τα εκτιμόμενα στοιχεία είναι αυτά τα οποία βρίσκονται ως στοιχεία στους ετήσιους λογαριασμούς. Και τώρα, με περισσότερη λεπτομέρεια από ό,τι στο παρελθόν, πράγμα το οποίο καταδεικνύει και τα όρια και τους περιορισμούς σε κάποιους τομείς διότι αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τη διάθεσή τους από τα κράτη-μέλη πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι πράγματι έγκαιρα διαθέσιμα. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βελτιώσει την αλυσίδα παροχής αυτών των πληροφοριών, πληροφοριακών στοιχείων. Αυτό επαρκεί όμως για να θεωρήσουμε ότι είναι πιο αξιόπιστες αυτές ε, οι ανακτήσεις. Ε. Είναι περισσότερο αξιόπιστο το θέμα αυτών των ανακτήσεων. Ε, τίθεται ένα ερώτημα αυτό. Δεν είναι μόνο θέμα επικρίσεων κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω πολύ καλή δουλειά κάνουν δεδομένων των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους. Όμως, στο τέλος τέλος, όταν έρχεται η ώρα να ληφθεί υπόψη αυτό το θέμα των διορθώσεων και των ανακτήσεων, αχρεωστήτων, αχρεωστήτως καταβληθέντων, υπάρχει ένα στοιχείο αβεβαιότητας όσον αφορά την διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία όλων αυτών των στοιχείων. Γι' αυτό θα απίθυνα έκκληση ή δυνατόν α ε, αναφέρεται στα θέματα εκτιμήσεων και ανακτήσεων και διορθώσεων θα πρέπει να βασίζεται στα σχέση με τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται. Κάποιος, ε, είναι η πρώτη φορά που ακούω τέτοια αριθμητικά μεγέθη, τέτοια στοιχεία καθ' όλη τη διάρκεια των ετών και δεν ήταν δυνατόν να αναφέρω τίποτα περισσότερο. Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία στους λογαριασμούς. Αυτά έχουν ελεγχθεί. Αυτά είναι τα ελεγμένα στοιχεία Αυτά είναι τα πιο αξιόπιστα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, μέσα στα συγκεκριμένα περιθώρια. Και θα έπρεπε να είμαστε πολύ σόφρονες και φρόνιμοι να μην παρεκκλίνουμε από αυτά. Τώρα, όσον αφορά και το κόστος ε, για τους ελέγχους ε, και τις δαπάνες σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί η Επιτροπή, είναι μία από τις μεγαλύτερες ελλείψεις που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δόθηκε επαρκής προσοχή, αγαπητοί συνάδελφοι, πόσο κοστίζουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, ποιες είναι οι δαπάνες τους. Και θα έπρεπε να επικαιροποιηθεί ή να μεταρρυθμιστεί κάποιο πρόγραμμα. Και αν είναι υπερβολικές οι δαπάνες, ε, τότε να μην πούμε «Α, είναι υπερβολικά δαπανηρό και δεν γίνεται τίποτα άλλο, οι δαπάνες πρέπει να καταβάλλονται με τον τρόπο αυτό». Πολλά μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί μια τέτοια κατάσταση και να πάμε καλύτερα. Αυτό το εγχείρημα λοιπόν όσον αφορά το κόστος των ελέγχων είναι πάρα πολύ σημαντικό input. Και φυσικά και το θέμα της απλούστευσης όταν έχουμε το θέμα της μεταρρύθμισης κανονισμών και διατάξεων υφισταμένων προγραμμάτων. Μετά έχω το επόμενο γράφημα ως διάγραμμα εδώ, το οποίο προσπαθεί να σας δώσει μια ιδέα για το τι πράγμα συζητούμε εδώ. Έχουμε ένα ποσοστό σφάλματος και υπάρχουν δύο σημεία πίεσης εδώ πρέπει να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος αφενός βελτιώνοντας ε, τους ε, μηχανισμούς και τα συστήματα ελέγχων τα ελεγκτικά συστήματα. Είναι ο μόνος τρόπος ε, για να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος. Βελτιώνοντας αυτό, αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά υποχρεωτικά περισσότερους ελέγχους. Συχνά σημαίνει καλύτερη εφαρμογή των υφισταμένων κανονισμών των ενισχύ ελέγχων. Και έχει επιδειχθεί αυτό, έχει αναφερθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να αποκομίσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ακόμα και από τους ενισχύ ελέγχους. Και υπάρχουν κάποιες διακοιμάσεις και παραλλαγές όσον αφορά τους ελέγχους και το κόστος και πρέπει να εξεταστούν. Υπάρχει πίεση όσον αφορά αυτό το στοιχείο. Άλλη πίεση προέρχεται από την άλλη πλευρά από την άλλη όχθη. Δηλαδή, βελτίωση του ποσοστού ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων. Η βελτίωση της ανάκτησης προέρχεται από την καλύτερη διαχείριση, σίγουρα, ουσιαστικά και η καλύτερη, από την καλύτερη εφαρμογή. Όχι μόνο για να έχουμε καλύτερα στοιχεία, πιο αξιόπιστα στοιχεία που θα μας διατίθενται, αλλά επίσης με το να διασφαλίζουμε ότι οι ανακτήσεις δεν θα είναι απλά κάποιες εντολές ε, ανάκτησης ποσών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα με τις ανακτήσεις που έχω είναι ότι έχουμε εντολές προς ανάκτηση που υπογράφονται, δηλαδή in the pipeline, εν ε, ε, εξελίξη δηλαδή, εν ρευστό, και την ε, ε, πραγματική ανάκτηση ποσών. Εμά αυτό που μα ενδιαφέρει δεν είναι η υπογραφή κάποια το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή ανάκτηση. Γιατί για ανάκτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ανάκτηση. Γιατί η μεν εξέλιξη με υπογραφή προς ε, εντολής δείχνει ότι έχουμε συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, αλλά το αποφασιστικό στοιχείο στο τέλο τέλο είναι να δούμε τις διάφορες εξελίξεις που μπορούν να ε, ε, συνεπάγονται όλα αυτά, δηλαδή προγράμματα τα οποία ίσως αποσύρονται ή ε, διαγράφονται και όλα αυτά να μπορούν να μπορούν να οδηγήσουν σε κατάργηση, άρση της εντολής ανάκτησης. Και εδώ λοιπόν υπάρχει αδυναμία στην αλυσίδα των πληροφοριακών στοιχείων. Να γνωρίζουμε δηλαδή περί τίνος πρόκειται, αλλά το τελικό ποσό είναι το σημαντικό αποτέλεσμα, το τελικό ποσό ανάκτησης. Αυτή η πίεση είναι που πρέπει να οδηγήσει στο να μειωθεί το χάσμα και να μειωθεί και ο κίνδυνος τελικά των αχρεωστήτων καταβληθέντων. Δεν είναι απλή αυτή η λύση, μια απλή εξίσωση, δεν μπορεί να γίνει μια νυχτή. Θα απαιτήσει χρόνο. Στην Γεωργία απέτησε πολύ χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιτευχθεί το θετικό αποτέλεσμα. Πήρε τουλάχιστον 6-7 χρόνια τουλάχιστον όταν ξεκίνησε η ε, μεταρρύθμιση, όταν τα συστήματα διαχείρισης άρχισαν να βελτιώνονται και στο τέλος τέλος κομμάτι-κομμάτι άρχισε να δίνει την τελική βελτίωση όπως ε, πρόσφατα. Λοιπόν δεν είναι ανέφικτο όταν ξεκινά κάτι δεν σημαίνει ότι για πάντα θα μένει έτσι όταν βλέπουμε ότι κάτι έχει με τον Α τρόπο θα πρέπει να το διαχειριζόμαστε και να το παρακολουθούμε ιδιαίτερα για κάποιους τομείς κινδύνου ή ευάλωτα σημεία ή υψηλή πίεσης και χώρες ιδιαίτερα ευάλωτες που πρέπει να ε, επικεντρωνόμαστε σε αυτά και σε αυτές. Και αυτό είπα, επικέντρωση και αξιολόγηση έγκαιρη αυτών των σημείων. Και μετά αυτό που κάναμε και αυτό βρίσκεται στην τάση, Αλλά αυτό που προσπαθήσαμε σε αυτό το έγγραφο να κάνουμε είναι να εξετάσουμε σε εξειδικευμένες εκθέσεις και αυτά τα στοιχεία και να δούμε ποια συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν και αυτό απορρέει συνήθως υπό την αποτελεσματικότητα των κριτηρίων οικονομικής διαχείρισης όπως αναφέρεται η συνθήκη και είναι και το αντικείμενο της ε, μεταρρύθμισης και αυτών των περιβόητων 20 εκθέσεων και αναφέρθηκε και αυτό και υπήρξε πίεση για να συζητηθούν όλα αυτά. Από όλε αυτές τις εκθέσεις τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να ανακεφαλαιώσουμε και να συνοψίσουμε εν περιλήψη τα κυριότερα στοιχεία και να επικεντρωθούμε κάπως σε αυτά. Προγράμματα δαπανών για παράδειγμα βρίσκουμε ότι δεν δίνουν εν γέννη αυτό το οποίο εμείς αποκαλούμε ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία. Και εδώ προτείνουμε να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή που θα δίνεται ίσως σε αυτή την προσέγγιση. Διότι στο τέλος τέλος τι συμβαίνει τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν είναι στοχεύουμε να υποκαταστήσουν τα εθνικά κονδύλια και χρηματοδότηση. Κάτι παραπάνω πρέπει να δίνουν και να παρέχουν. Να παρέχουν ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία. Αυτό δεν είναι. Ε, αυτό πρέπει να αντανακλάται λοιπόν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό πρέπει να καθοριστεί επακριβέστερα και τα νέα προγράμματα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό το στοιχείο. Είναι μείζον εγχείρημα αυτό. Δεν είναι ε, μικρό υπόθεση και πρέπει να δοθεί αναγκαία προσοχή. Είναι πολύ απαιτητική υπόθεση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Ευρωβουλή και το Συμβούλιο να υπάρξει επαναπροσανατολισμό επ' αυτού, μια νέα κατεύθυνση, νέα προσέγγιση. Γι' αυτό το εντάξαμε σε αυτό το πλαίσιο. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι πολλέ πολλές φορές από του στόχου των προγραμμάτων είναι ευρύτατοι, ασαφεί και πολλές φορές ε, αλληλοσυγκρουόμενοι. Και πάλι στο τέλο τέλο, όταν καταλήγουμε στο να συγκρίνουμε αυτού του στόχου για να δούμε αν επιτέχθηκαν, επιτέχθησαν τα αποτελέσματα. Καμιά φορά λέμε, μα γιατί αυτό καθορίστηκε με αυτόν τον τρόπο ο στόχος. Δεν είναι εφικτό να επιτελεστεί με τον τρόπο αυτό ως προσέγγιση. Τώρα, και όσον αφορά και την ε, διασύνδεση όλων αυτών των προσπαθειών προς ένα τελικό στόχο και υπερβολική, υπερβολικά περίπλοκα ε, κριτήρια για την επιλεξιμότητα. Αναφερθήκαμε σε αυτά τα θέματα σε ειδικέ εκθέσεις όπου σημειώσαμε κάποια πράγματα. Τώρα, μη σαφή ρόλοι, ασαφή ρόλη και ασαφή προσδιορισμός ευθυνών, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινή ευθύνη για τη διαχείριση, ελλείψει όσον αφορά την παρακολούθηση και αξιολόγηση ανεπαρκής πρόσβαση σε στοιχεία και έγγραφα, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινή διαχείριση και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και φορέων. Τι μπορεί παραπάνω να γίνει και θέλω να ολοκληρώσω για να μην μακρηγορήσω υπερβολικά. Ο περαιτέρω προβληματισμός για αυτή την ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία που προανέφερα. Νομίζω η Ευρωβουλή θα έπρεπε πραγματικά ίσως να το εξετάσει αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή αρχή προς ανατολισμού. Γνωρίζω από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον πρόεδρο Μπαρόζο και από τα έσω έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα ότι είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο αυτό που μπορεί να ακολουθηθεί όταν σχεδιάζουμε παρεμβάσεις ε, και σε σχέση με το στόχο της αφήνεια των στόχων, την διαφάνεια, την, ε, το εφικτό των στόχων και την λογοδοσία απλή όρη πολλές φορές, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν ε, προσεγγίζονται με τον πιο σωστό τρόπο. Και φυσικά η εξάντε αξιολόγηση και η αξιολόγηση επιπτώσεων που πρέπει να ενδυναμωθούν περαιτέρω. Εν γέννη αυτό το οποίο γενικά απαιτεί η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι συχνά πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο εξειδικευμένο από αυτά τα οποία απαιτούν οι εθνικές αρχές από πλευράς τους. Λοιπόν, γεγονός όμως παραμένει ότι αντιμετωπίζουμε κονδύλια ευρωπαϊκά εδώ τα οποία διατίθενται. Και αυτές οι πτυχές, αυτή η πτυχή είναι πάρα πολύ σημαντική θα έλεγα και θα έπρεπε να ενδυναμωθεί. Η δημοσιονομική αναθεώρηση θα έπρεπε να ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα να ληφθούν υπόψη προετοιμάζοντας ένα νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι δεν είναι. Και σε σχέση και με τη βελτίωση, όπως είπαμε, για τις ε, δαπάνες ε, και τον όγκο δαπανών, όσον αφορά την ποιότητά τους, βελτίωση. Και όσον αφορά και τα input-output και με αυτά που ακούσαμε από την Επιτροπή εχθές και την τελευταία φορά που έγινε παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς αυτή την κατεύθυνση προβληματίζονται στην Επιτροπή, θα έλεγα, με σοβαρό τρόπο. Και αυτό κιόλας είναι μια διαφορετική αρχή προσανατολισμού. Είναι κάτι διαφορετικό από το να επικεντρώνεται κανείς σε ε, ε, λογαριασμούς ε, και απλά έγγραφα καταβολών ποσών και πληρωμών. Να δει κανείς το εύλογο ύψος δαπανών που πρέπει να επιτευχθεί. Smart regulation, ευφυής νομοθεσία και ευφυής διατάξεις που πρέπει να δημιουργηθούν. Όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον πρόεδρο Μπαρόζο σε παρέμβασή του. Χρειαζόμαστε ευφύ παρέμβαση νομοθετικά και σε δια... αφορά διατάξεις και ρήτρε. Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να βελτιωθούμε όσον αφορά την έννοια του ανεκτού ποσοστού σφάλματος. Να δούμε το κόστος και το όφελος. Πού βρισκόμαστε δηλαδή και το επόμενο βήμα θα είναι το τι πρέπει να γίνει υποχρεωτικά ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε προς ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ κόστους δαπανών και ωφέλου, ώστε να μην δαπανώνται, να μην διασπαθίζονται τα κονδύλια ή να μην πηγαίνουν στράφοι και τα ωφέλη από αυτούς τους ε, ελέγχους ε, να είναι δεδομένα με καλύτερο input και καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτά εν αγαπητοί συνάδελφοι είναι μια σύνοψη του πολύ συντόμου αυτού εγγράφου που προετοιμάσαμε από πλευρά ε, της Επιτροπής για την Επιτροπή και θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι θετικές αρχές ανατολισμού σε σχέση με τη νέα Επιτροπή και τη νέα εντολή της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρέσλε έχει ζητήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπονίτσι. Είναι, ας το πω έτσι, θα έλεγα, μία από τις τελευταίες σας παραστάσεις εδώ θα έλεγα. Δυστυχώς ε, δεν θα ε, συνεχίσει η θητεία σας. Λυπάμαι γιατί σας κοστάμε πάρα πολλά θετικά και ξεκινώ με θερμές ευχαριστίες προς εμάς, διότι καταφέρατε τις αιτήσει εκθέσεις να τις κάνετε πιο εύληκτες, πιο κατανοητές. Και επειδή μας ανοίξατε τα μάτια και αποκαλύψατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε σχέση με τη διαχείριση των κονδυλίων του προϋπολογισμού και σας ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά. Θα ήθελα κάποιες ερωτήσεις να σας διατυπώσω. Εχθές είχαμε αυτή τη σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Διευθυντή για τα Περιφερειακά. Ποιο είναι το ποσό τώρα των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Αν θυμάμαι σωστά στην σημείωση 2000, για το 2008 λέει ε, τόσα δισεκατομμύρια ευρώ αν θυμάμαι καλά για τα διαθετικά ταμεία. Θα ήταν σημαντικό για μας ως Ευρωκοινοβούλιο να υπάρξει ποσό, να αναφέρεται ένα συγκεκριμένο ποσό και ένα ποσό για την ανάκτηση αχρεωστήτως ε, καταβληθέντων. Ποιο είναι αυτό το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθέντων και των ανακτήσεων από τα αχρεωστήτων καταβληθέντα. Θα μας ενδιαφέρει αυτό. Να έχουμε μια τέτοια, ένα τέτοιο πίνακα, να μπορούμε να συγκρίνουμε σε σχέση π.χ. με το 2008. Τα στατιστικά στοιχεία από το 2000 έως το 2006 έχω εξοικειωθεί με αυτά και εξαρτάται τι βλέπει κανεί και τι μετρά και ποιον ρωτά για τι απαντήσει που παίρνει. Να δούμε το πώ θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτά τα συστήματα. Σημαντικό αυτό. Όσο περισσότερο ασχολούμαι με αυτό το θέμα, τόσο περισσότερο καταλήγω στο συμπέρασμα ότι οι δικέ μα αντιφάσει και οι αντιφάσει του Συμβουλίου είναι οι κύριε υπεύθυνε για μια κατάσταση που εδώ και πέντε χρόνια τώρα συζητάμε ότι πρέπει να σημειωθούν πρόοδοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να συζητάμε όταν, για ένα σύστημα βελτίωσης όταν έχουμε την ε, ε, περίπτωση της Βουλγαρίας. Ποτέ δεν πάγωσαν περισσότερο από ένα μικρό ποσοστό των κονδυλίων προς τη Βουλγαρία παρόλη την αρνητική κατάσταση των πραγμάτων. Ένα σύστημα το οποίο δεν θέτει η σημασία στο να υπάρχουν κυρώσεις εις βάρος των κρατών μελών που δεν ευθυγραμμίζονται είναι ένα άχρηστο σύστημα. Γιατί διαιωνίζονται τα προβλήματα και κάθε χρόνο πάμε με το καρότσι τα λεφτά στις χώρες αυτές και τους τα διαθέτουμε. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Επειδή ουσιαστικά ποτέ δεν είμαστε αρκετά στεναροί και αποφασιστικοί ώστε να τερματιστούν αυτέ οι καταστάσει. Ποτέ δεν είδαν να υπάρχουν κυρώσει σε αυτά τα κράτη. Και βλέπουμε και στην Ελλάδα τώρα την απουσία στεναρότητα και συνέπεια στι δράσει μα. Θα με ενδιαφέρε πώ το βλέπετε εσεί. Τι μπορούμε να κάνουμε ω προ αυτά. Με ενδιαφέρον σημείωσα και έλαβα υπόψη ότι τι ειδικέ εκθέσει όσον αφορά και το, την ετήσια έκθεση τα συνδέεται αυτά μέσα σε αυτό το πλαίσιο και στο έγγραφο αυτό είναι ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Όμως δεν είμαι πρόθυμη αγαπητοί συνάδελφοι να περάσω τα επόμενα πέντε χρόνια με αυτό το οποίο έκανα τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Να διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς και μετά να μην γίνεται τίποτα και να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος. Α, και ο κύριος Λιμπεράτσκι έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Μετά από την παρουσίαση την οποία έκανε ο κύριος Μπονίτσι, μου έχει δημιουργηθεί μια μικρή σύγχυση. Όταν κάποιος φεύγει από τη θέση του, ε, φυσικά αφήνει ένα κενό, αλλά είναι κρίμα που φεύγετε εσείς Αν παρακολούθησα καλά την παρουσίασή σας, είπατε το εξής. Περιμένετε λίγο περισσότερο για την απαλλαγή. Περιμένετε ένα πιο ξεκάθαρο πρόγραμμα της Επιτροπής και μετά να αποφασίσετε την απαλλαγή. Κατάλαβα καλά, κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε κύριε Μπονίτση είναι το κληροδότημα που απορρέει από ερωτήσεις και πέρα από ερωτήσεις επιπλέον θα έλεγα ε, προσπάθειες ε, συνολικά βελτιώσεων διότι επί παντός του επιστητού, διότι να δούμε ποια είναι η πρόσθετη αξία των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να αναδιαβιβάσω το ερώτημα. Εσείς αξιολογήσατε ποια είναι αυτή η πρόσθετη αξία και είπατε δεν υπάρχει μεγάλη πρόσθετη αξία. Ε, ποια είναι λοιπόν για σας η πρόσθετη αξία, διότι δουλεύουμε όλα τα θεσμικά όργανα προσπαθώντας ακριβώς να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πρόσθετη αξία σε όλες τις πολιτικές και στις μεταφορές για παράδειγμα. Είδαμε και τις διαμεθοριακές πτυχές διασυνοριακά. Ένα κράτος το οποίο επενδύει για παράδειγμα εδώ και όχι αλλού ε, όσον αφορά τις, ε, τα σύνορα. Αυτό το οποίο θέτετε εσείς είναι μία από τις θεμελιώδεις πτυχές για το μέλλον και το, στο μέλλον θα είναι όλο και πιο σημαντικές όταν έχουμε και το θέμα επανεθνικοποίησης πολλών πολιτικών και της πολιτικής συνοχής και θα δούμε τα αποτελέσματα στο μέλλον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω από τη σοφία σας και την πείρα σας με αυτό το κληροδότημα ποια θα ήταν, μπορείτε να εμβαθύνετε περισσότερο σε αυτά τα στοιχεία αυτή η πρόσθετη αξία, ποια θα ήταν για αυτή την πρόσθετη αξία που θα είναι η λιδία λίθος για το μέλλον για μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Γκέιρ. Πρώτα θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου στις ευχαριστίες των συναδέλφων προς εμάς κύριε καθηγητά Μπονίτσι. Λυπάμαι και εγώ για το ότι θα μας εγκαταλείψετε. Μπορώ και προσωπικά ο ίδιος να σας πω, αλλά και για την ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών να σας πω ότι ακόμα και στο μέλλον όταν δεν θα έχετε αυτό το αξίωμα στο μέλλον θα χρειαστούμε να χρησιμοποιήσουμε τις συμβουλές σας και θα προσφύγουμε, θα προστρέξουμε σε εσά. και ένα προσωπικό εδώ αν θέλετε ε, σχόλιο έχω και ένα μικρό μουσείο παραθεμάτων αν θέλει κανείς μεταφορικά να περιγράψει κάποιο πρόβλημα να δει τη δική σας ε, ε, πρόταση ως παράθεμα. Η απλούστευση είναι δύσκολο εγχείρημα είπατε. Εγγράφετε αυτό το παράθεμά σας στο μουσείο μου, μουσείο μου παραθεμάτων. Θα ήθελα εδώ αμέσω άρρηκτα να συνεχίσω και να πω κάτι. Αυτό η μείωση του ποσοστού σφάλματος που είναι ένα θέμα για να, που για να το πετύχουμε αγωνιζόμαστε σκληρά. Εδώ διτά το αντιμετωπίζουμε. Αφενός μείωση του ποσοστού σφάλματος. Εδώ θα μπορούσε η απλούστευση να είναι μια προσέγγιση εφικτή. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και την αύξηση του ποσοστού ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων. Ρώτησε συνάδελφος πιο πριν και δεν χρειάζεται χρειάζεται να επαναλάβω εγώ την ερώτηση που έκανε. Όμως, τούτων λεχθέντων, εγώ θα ενδιαφερόμουν πάρα πολύ μέσα σε αυτόν τον κύκλο να μας λέγατε ποιες είναι οι σκέψεις σας στον τομέα της απλούστευσης, ιδίως στο output, να μας πείτε τι σκέφτεσαι σχετικά. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο πάλι στον κύριο Μπονίτσι για να κλείσει. τέθηκαν αρκετές και δύσκολες ερωτήσεις. Ανάκτηση ποσών. Πόσα χρήματα δόθηκαν ενώ δεν θα έπρεπε να δοθούν. Περίπλοκη ερώτηση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο έτος, να δούμε το τελικό αποτέλεσμα, να εκτιμήσουμε την δημοσιονομική επίπτωση και να προβάλλουμε την, να κάνουμε μία προβολή στο σύνολο της χρονικής περίοδου. Αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός χρόνου. Βέβαια πολλά προγράμματα είναι πολυετή και μερικές φορές αναγκαζόμαστε να κάνουμε διορθώσεις σε ιστερότερες φάσεις. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Και γι' αυτό απαιτούμε πληροφορίες αν θέλετε και χρειαζόμαστε τις πληροφορίες για ανακτήσεις ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα. Ο πολιετής χαρακτήρας επηρεάζει θα έλεγα και καθιστά την κατανόηση ορισμένων επενδύσεων, ορισμένων μάλλον καταβολών, ε, δύσκολη να κατανοηθεί. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε για αρκετά εκατομμύρια τα οποία θα μπορούσαν να ανακτηθούν. Δεν έχω τους πίνακες όλους αναλυτικά, αλλά για το 2009 στον τομέα της συνοχής μιλάμε για 900 εκατομμύρια, τα οποία ελέγξαμε. Ακούμε βέβαια στοιχεία και πληροφορίες μερικές φορές για δις εκατομμύρια ποσά ευρώ, αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τέτοιους αριθμούς. Να θυμηθείτε παρακαλώ ότι όταν λέμε την λέξη τουλάχιστον, το at least στα αγγλικά, αυτό αν θέλετε είναι το τέλος μιας στατιστικής προβολής. Το συνολικό ποσό, το μέσο ποσό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από αυτό στο οποίο καταλήγουμε. Το να προσπαθήσουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε εμείς το άκρον μια στατιστικής προβολής στο σύνολο του πεδίου που θέλουμε να καλύπτουμε δεν είναι ιδιαίτερα σοφό. Και γι' αυτό ακριβώς το ελεγκτικό συνέδριο λέει συνέχεια τουλάχιστον, τουλάχιστον 11% στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ελέγξαμε 26 δις σαν παράδειγμα το προηγούμενο έτος στον τομέα της συνοχής. αν θέλουμε να αξιολογήσουμε απόλυτα τα συγκεκριμένα ποσά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια διαφορετικού τύπου αναλυτική μορφή ελέγχου των λογαριασμών. Νομίζω ότι απαιτείται, εν πάση περιπτώσει, μια πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία, η οποία θέλει περισσότερο χρόνο και δεν μπορώ να σας πω τόσο, δεν μπορώ να σας πω 2,6 δις σαν παράδειγμα. Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο τίποτα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα ανακτηθέντα ποσά και τον πολυετή χαρακτήρα και ίσως αυτό να καταλήξει σε περισσότερα, σε μεγαλύτερα ποσά από αυτά τα οποία έχουμε εκτιμήσει. Είμαστε όμως ιδιαίτερα επιφυλακτικοί να ποσοστικοποιήσουμε αν θέλετε τις μελέτες αυτές που έχουμε κάνει. Υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι τεχνικοί λόγοι που δεν μου επιτρέπουν να σας δώσω ένα αριθμό σε ευρώ. Πάντως το θέμα είναι ένα. Έχουν δοθεί χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί. Δεν ξέρουμε πόσα είναι, δεν ξέρουμε πού ακριβώς. Δεν ξέρουμε αν οι προηγούμενες περίοδοι για τις οποίες εκ των υστέρων έχουμε περισσότερα στοιχεία αποτελούν ένα παράδειγμα το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς στους πίνακες που παρουσίασα αναφέρθηκα στην πίεση που προέρχεται ε, από κάτω προς τα πάνω σχετικά με την ανάκτηση αχρεωστήτων σκαταβληθέντων ποσών. Λέμε τουλάχιστον επαναλαμβάνω 11%. Και αυτό το 11% δείχνει σαφέστατα ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το οποίο έθεσε σαν ερώτημα ο κύριος Λιμπεράτσκι, εσείς θα πρέπει να το σταθμίσετε και να το αποφασίσετε. Φέτος υπήρξαν βελτιώσεις σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και σε σχέση με τον προπροηγούμενο και πάει Αυτές οι βελτιώσεις κρίνονται επαρκείς. Μπορεί κανείς να εκφράσει διάφορες απόψεις επ' αυτού. Η δική μου αντίδραση είναι να πω ότι υπήρξαν από τι πιο σημαντικές αλλαγές στα αποτελέσματα. Και αυτό το θεωρώ θετική εξέλιξη. Το ερώτημα είναι θα πρέπει κανείς να πει να συνεχίσουμε σε μια προσπάθεια και άλλων βελτιώσεων ή ίσως πρέπει να ζητήσουμε ένα σχεδιασμό για το πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση για κάποια χρόνια. Εάν νομίζουμε ότι περιμένοντας μέχρι τέλος του έτους θα προκύψει μια λύση, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Η λύση είναι πολυσχηδής, είναι περίπλοκη, απαιτεί την συμμετοχή των 27 χωρών μελών, ίσως και περισσότερων σύντομα, χρειάζεται κοινή διαχείριση και μια κατάσταση και έρχομαι σε αυτό που είπε ο Σκάιερ ότι είναι δύσκολη η απλοποίηση ζήτησα από τον Επίτροπο Κάλλας γιατί άραγε δεν μπορούν να απλοποιήσουν περισσότερο τους κανόνες της έρευνας στα πανεπιστήμια. Και είχα όταν ήμουν υπουργό. Είχα μια επιτροπή η οποία έκανε κάποιες προτάσεις, είχε όμως και την εξουσία να αποφασίζει. Στο στήθμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλλάζει βέβαια τώρα αυτό. Μπορεί κανείς να προβάλλει μια αξίωση για overheads. Θα δούμε τι εννοεί. Αυτά μπορεί να είναι με χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά βλέπεις ότι ο κανονισμός λέει ότι τα overheads πρέπει να έχουν σχέση με το πρόγραμμα έρευνας. Άμα όμως έρχεται κάποιος και λέει ότι για αυτά τα overheads, τα επιπλέον, το επιπλέον κόστος δηλαδή εν τέλει, χρειαζόμαστε παραπάνω από τα 10.000 ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά, ε, τότε χρειαζόμαστε άλλο ειδικό, ε, ειδική πρόβλεψη για να μπορεί να προβλέπει αυτή την έξτρα παραπάνω χρηματοδότηση. εν τέλει κάποτε καταλήγετε να δώσετε περισσότερα στη βάση τιμολογίων, άλλες φορές λιγότερο. Αυτό που μου είπε ο Επίτροπος Κάρας είναι ότι κοιτάξτε τώρα τότε θα πάμε στο Συμβούλιο, στο Υπουργών και θα, και θα πούμε ότι το κόστος έρευνας στο τάδε πανεπιστήμιο, στην τάδε χώρα και μετά στο άλλο πανεπιστήμιο της άλλης χώρας δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε benchmark επομένως. Το ένα έχει υψηλότερο κόστος, το άλλο έχει χαμηλότερο κόστος. Και αντί να προσπαθήσουμε να βάλουμε δύο μέσους όρους, ένα για υψηλό κόστος, ένα για μέσους κόστος, για, μέσο, για χαμηλό κόστος, ε, τότε θα πούμε όχι, μόνο τιμολόγια. Όσα τιμολόγια υποβάλλονται, αυτά πληρώνονται. Αυτό ανοίγει μια πόρτα εν τέλει για παραβίαση των κανονισμών. Και επομένως μπαίνουμε τελικά σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή θεσπίζονται οι κανονισμοί, πάμε, ελέγχουμε και βλέπουμε ότι παραβιάζονται. Δεν ακολουθούνται. Αυτό αποτελεί απάτη στις περισσότερες περιπτώσεις. Όχι. Γιατί αν έχουμε υποψία για απάτη, στέλνουμε την υπόθεση στην Όλαφ. Από την άλλη μεριά, είναι καλό να υπάρχουν τέτοιε περιπτώσεις. Όχι. Γιατί προκαλούνται και υπερβολέ. Γίνονται αδικαιολόγητες, προβάλλονται αδικαιολόγητες αξιώσεις. Και επειδή οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα επινοητικοί, δεν είναι δύσκολο να σκεφτούν ορισμένοι τρόπους για να μεγιστοποιήσουν τα όσα απολαμβάνουν, τα όσα βάζουν στην τσέπη δηλαδή από τα ταμεία αυτά. Αυτό κάνουν. Δεν τους κατηγορώ απαραίτητα. Όμως προκαλεί προβλήματα και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου λόγω της έλλειψης διαφάνειας, λόγω της έλλειψης θετικού μηνύματος σε ορισμένους σημαντικούς τομείς, αυτά ερμηνεύονται ως κατασπατάληση χρήματος. Μπορεί και να είναι, διότι γίνονται έλεγχοι οι οποίοι τελικώς δεν οδηγούν σε δυσκολίες. Και στο επίπεδο του Συμβουλίου λοιπόν η προσπάθεια απλοποίησης γίνεται εν τέλει μια ακροβασία που εν τέλει ανακόπτει την πρόοδο πολλών προτάσεων που θα μπορούσαν να βελτιώσουν κάποιες καταστάσεις το τελικό τους αποτέλεσμα. Και έρχομαι στο τελευταίο. Για την πλευρά της, των εκροών του output. Γιατί, συγγνώμη, οι δικές μας εκθέσεις είναι σημαντικές διότι ρίχνουν ιδιαίτερη δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία, στην αποτελεσματικότητα, στην αποδοτικότητα. Δηλαδή, επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί. Αυτό που προτείνουμε είναι να γίνει ένας επαναπροσανατολισμός στις δημοσιονομικές ρυθμίσεις, όπου αντί να ρίχνετε το βάρος σε τιμολόγια και σε ποσοστά επιτρεπόμενων εξόδων και τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Να ρίξουμε βάρος κυρίως στο ποθητό αποτέλεσμα και να υπάρξει ένας τρόπος να αξιολογηθεί αυτό το αποτέλεσμα και να καθορίσει ένα ποσό, η Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα, για να πει ότι το project μου κόστησε 10 εκατομμύρια ευρώ, γι' αυτό το μερίδιο της Ένωσης θα πρέπει να είναι 6 εκατομμύρια να γίνει και μια σωστή διαδικασία προσκλήσεως ενδιαφέροντος κτλ. Και αν κοστίσει παραπάνω τότε θα πρέπει η χώρα μέλος να αναλάβει. Να ασκηθεί λοιπόν κάποια πίεση στις αρμόδιες αρχές ώστε να μην ξεπεράσουν το κόστος αυτό. Εάν το project τελικά κοστίσει λιγότερο, αλλά πόσα project κοστίζουν λιγότερο. Μου τύχανε ένα-δυο. Αλλά μέσα στις εκατοντάδες project που έχω δει, ίσως να έχουμε και χίλιες και χίλιες τρακόσες τέτοιου είδους συναλλαγές κάθε χρόνο. Σπάνια, ε, να είδα μία φορά σε όλες αυτές να είδα μια υποτίμηση, δηλαδή να κόστησε εν τέλει λιγότερο. Αυτό χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, αλλά μέχρι ενό σημείου. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να επανεξεταστούν όλες οι διατάξεις μας, οι κανονισμοί μας. Υπάρχει βέβαια αντίσταση στην αλλαγή από διάφορες πλευρές και λόγω τη απέτηση πρώτα να υποβάλλεται πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την εξετάζει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και είναι μακρόχρονη αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό καμιά φορά πρέπει να γίνεται με επίγοντα χαρακτήρα, ώστε στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με διαφορετική πρόπτικη. Η λύση δεν είναι απλή και ούτε μπορεί να γίνει με το γύρισμα ενός διακόπτη. Νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Νομίζω ότι είναι δυνατό να επανεξεταστούν ένα πράγμα που σημείωσα χθε. Είναι ότι δίνεται σωστά έμφαση στη νέα περίοδο προγραμματισμού στα διαρθρωτικά ταμεία. Και καλέμε εκεί better regulation και ελπίζουμε να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε πότε γιατί είναι αργή η διαδικασία. Αλλά τι γίνεται με τις τρέχουσες πληρωμές για την τελευταία περίοδο προγραμματισμού. Μπορεί να γίνει κάτι για να διορθωθούν αυτά γιατί το ποσοστό σφάλματος για φέτος θα βασιστεί κατά δύο τρίτα τουλάχιστον για την συνοχή στην τελευταία περίοδο προγραμματισμού. Και εκεί μπαίνουν οι αιτήσεις εκθέσεις και το management και ίσως να μην υπάρχουν επαρκείς πόροι για την διαχείριση της περιπλοκότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα αυτά τα προγράμματα. Νομίζω είναι 500 επιχειρησιακά προγράμματα σε 27 χώρες μέλη και σε όλες τις περιφέρειες. Είναι περίπλοκο, πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι μπορεί να αντιμετωπίσει οποτεδήποτε κάποια μία χώρα μέλος. Ίσως λοιπόν χρειάζεται να υποστηριχθούν και οι προσπάθειες της Κομισιόν να βελτιώσει τους πόρους της ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα. Εμείς ως δικαστήριο έχουμε μεγάλη δυσκολία να κάνουμε περισσότερα μία από τις διαρκείς συζητήσεις που κάνω με τους συναδέλφους μου, δεν είναι μυστικό αυτό, είναι αν δεν θα ήταν πιο σωστό να χωριστεί η συνοχή σε δύο, κοινωνικό ταμείο και περιφερειακό ταμείο. Στην δική μας ανάλυση έχουμε ένα δείγμα. Δεν θα ήταν καλύτερα η ανάπτυξη υπεύθυνο ξεχωριστή από την αγροτική οικονομία. Να αυξηθεί επομένως το υποδείγμα για την ε, ανάπτυξη τη που δεν θα είναι ανεξάρτητο, θα μας προσφέρει όμως περισσότερες πληροφορίες για αυτό το υπό σύνολο και το πώς θα αντιμετωπίσουμε την έρευνα. Μήπως πρέπει να είναι από μόνη της. Αυτά είναι διάφορα στοιχεία. Η κυρία Σαντάλοβα είναι παρούσα για να μιλήσει για τους οργανισμούς. Α, οι οργανισμοί, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τόσους πολλούς οργανισμούς και είναι τεράστια πρόκληση να αντιμετωπίσει κανεί όλα τα προβλήματα των οργανισμών και να μπει στου λογαριασμού του με κάποια ε, λεπτομέρεια. Όταν ζητούμε πόρους, έχουμε περιορισμένους πόρους. Ένα άλλο τομέα τομέας, με τον οποίο και θα κλείσω, είναι αυτό το νέο project για τα πιλωτικά προγράμματα. Τι κάνουμε. Έχουμε τέσσερις χώρες μέλη που υποβάλλουν εθνικές δηλώσεις. Πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές. Υπάρχει και, πρόβλημα χρονισμού, πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα, και πρόβλημα μεθοδολογίας. Καταλήξαμε σε ένα κόνσεπτ κοινών ελέγχων, ώστε συμφωνήσαμε με τρεις χώρες μέλη, δύο από τις οποίες κάνουν εθνικές δηλώσεις. Όταν κάνουν την αναλυσή τους οι χώρες αυτές, εμείς συμμετέχουμε Παίρνουμε δηλαδή και εμείς από τις δικές μας DAS στοιχεία και οι πληροφορίε που χρησιμοποιούν για τη δική τους εθνική δήλωση και που τις χρησιμοποιούν ανεξάρτητα από μας και αυτόνομα, έχουμε και εμείς καλύτερες πληροφορίε για αυτά, κάτι που καθιστά και τη δική μας τη ζωή πιο εύκολη, να μπορούμε δηλαδή να αξιολογήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα αυτά. Νέα εξέλιξη βέβαια αυτή συμμετέσχαμε και σε ελέγχους απόδοσης μαζί με εθνικούς οργανισμούς, όχι ποτέ όμως στην σύνταξη των DAS. Αυτό είναι pilot project. Έχουμε και έναν άλλο αριθμό χωρών μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν, που δεν μπορέσαμε όμως να πετύχουμε τη συνεργασία αυτή λόγω έλλειψης πόρων και είπαμε ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε παραπέρα το concept αυτό των συνεργασιών με την τεχνογνωσία των χωρών μελών και τη δική μας τεχνογνωσία. Αυτά σας ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 21 της ημερήσιας διάταξης απαλλαγή για το 2008. Έλεγχος των εξαρτημένων οργανισμών. Κυρία Ματιώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση ταχύτατα και μετά δεν θα αναφερθώ στις 26 υπηρεσίες αλλά σε κάποια παραδείγματα. Τρία βασικά θέματα. Το πρώτο αφορά τα εγκάρσια προβλήματα θα έλεγα τα οποία αφορούν πολλές από αυτές τις υπηρεσίες μεταφορές και ακυρώσεις ε, λειτουργικών δαπανών. Είναι μια διαπίστωση σε πάρα πολλά από τα όργανα αυτά, από τους οργανισμούς αυτούς. Κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές δυσκολεύονται να διαχειριστούν μια σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού τους. Αυτή η διαπίστωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά από το Κοινοβούλιο σαν αρχή επί του προϋπολογισμού τα μέλη μέσω των ψηφοφοριών για τον προϋπολογισμό επηρεάζουν άμεσα. Και αναφέρομαι εδώ στην αρχή την Ευρωπαϊκή για την ασφάλεια των τροφίμων, την πρόληψη των ασθενειών, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Frontex, την Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στους χώρους εργασίας και για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την βελτίωση ε, των συνθήκων εργασίας και για το ε, όργανο ή οργανισμό Eurojust. Το πρόβλημα επίσης ε, των προμηθειών είναι ένα σαφέστατο πρόβλημα ιδιαίτερα στα παλαιότερα όργανα, στους παλαιότερους οργανισμούς οι οποίοι οι οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις συστάσεις οι οποίες τους γίνονται στον τομέα αυτό. ΣΕΙΠΟΛ, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Δικτύων, Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Υπηρεσία και Eurofund. Το θέμα του ανθρώπινου δυναμικού είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Από την ποιότητα των προσλήψεων εξαρτάται ουσιαστικά η ποιότητα εργασίας μιας τέτοιας υπηρεσίας και οι προσδοκίες που έχουμε από μια τέτοια υπηρεσία. Δυστυχώς ασκούνται πάρα πολύ σοβαρές κριτικές από το ελεγκτικό συνέδριο σχετικά με ανεπάρκειες γύρω από τον προγραμματισμό και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού δεν είναι δυνατό να γίνει δεκτό σήμερα να βλέπουμε σε κομβικά σημεία του οργανογράμματος συμβασιούχους υπαλλήλους, ιδιαίτερα στον, στον οικονομικό τομέα και να υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για τις ε, διαδικασίες πρόσληψης. Θυμίζω επίσης ότι πολλές από τις υπηρεσίες αυτές δεν έχουν συνάψει συμφωνίε έδρας με τις χώρες υποδοχής και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Τρίτον, παρατηρήσεις για το σύστημα λειτουργίας. Το εσωτερικό ελεγκτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σαν στόχο να κάνει συστάσεις στις υπηρεσίες αυτές για να διορθώνονται οι ελλείψεις στις οποίες αναφέρθηκα. Θα ήθελα να υπάρξει λίγη ησυχία γιατί ο θόρυβος με ενοχλεί. Είναι απαραίτητο οι συστάσεις να μην αγνοούνται από τους διευθυντές των υπηρεσιών αυτών και από τα διοικητικά του συμβούλια. Σε κάθε μία από τις εκθέσεις αναφέρομαι στις εσωτερικές ελεγκτικές διαδικασίες, αναφέρομαι στις πληροφορίες που δίδουν οι υπηρεσίες αυτές σχετικά με το είδος της ενημέρωσης και όλα αυτά θα επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να κατανοήσουν σωστά τον ρόλο που παίζουν τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου. Πειθαρχικές διαδικασίες. Θα ήθελα να συγκεκριμενοποιείτε ιδέα ενός κοινού πειθαρχικού συμβουλίου που θα παραπέμπει μετά από έρευνα της ΟΛΑΦ στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα πρέπει να ξεκινήσει ε, μια συντονισμένη επικοινωνία ανάμεσα ε, στις υπηρεσίες των οργάνων αυτών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της πειθαρχίας, για τον σεβασμό μάλλον της πειθαρχίας. Αυτό βέβαια αφορά και τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλουμε να υπάρξει σημαντική πρόοδος σε τομείς που αφορούν τη δική μας Επιτροπή, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν σε επίπεδο διοικητικού πολιτισμού σε εισαγωγικά και κυρίως σε επίπεδο πρόσληψης του Διευθυντή. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και είναι ανεξάρτητες οι υπηρεσίες αυτές, έχουν πάντα μια γενική διεύθυνση αναφοράς, η οποία θα πρέπει διοικητικά να τις βοηθά. Αυτό δεν γίνεται με ομοιογενή τρόπο σε όλες τις γενικές διευθύνσεις και γι' αυτό ο συντονισμός είναι απαραίτητος ιδιαίτερα για τις πολύ μικρές υπηρεσίες. Διοργανικός διάλογος. Πολλά από τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται από την ομάδα εργασίας στη διοργανική για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Οι, τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία και τα ευρωπαϊκά όργανα θα έπρεπε να περιμένουν το τέλος των εργασιών αυτής της ομάδας πριν προτείνουν τη δημιουργία νέων υπηρεσιών. Έτσι, λυπάμαι για τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 1η Φεβρουαρίου 2010 που ε, θα έχει σαν στόχο τη δημιουργία μιας υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την επεξεργασία των λιμάτων, των αποβλήτων, συγγνώμη. Είναι σαφές ότι πρέπει να περιμένει κανείς ε, μια στενή συνεργασία ανάμεσα στις υπηρεσίες αυτές. Πολλές φορές θα μπορούσαμε να προτείνουμε και συγχωνεύσεις ανάμεσα στις υπηρεσίες αυτές και τη διοικητική του συνεργασία στα πλαίσια μια σωστή δημοσιονομικής λειτουργία. Τίθεται το θέμα εδώ και το θέμα του μεγέθους, θα έλεγα, του Διοικητικού Συμβουλίου των εκπροσώπων που, που, αποτελούν, που συνιστούν τα Διοικητικά Συμβούλια, κάτι το οποίο για τις μικρές υπηρεσίες ε, αντιπροσωπεύει ένα πάρα πολύ σημαντικό κόστος. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Αστυνομία και η Υπηρεσία για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας που έχουν περισσότερα μέλη στο διοικητικό του συμβούλιο από ό,τι έχουν εργαζομένους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίζει πιο σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να μην δημιουργείται ε, μια μειοψηφία η οποία κάθε φορά να μπλοκάρει και να παγώνει τις εργασίες. Τώρα, επιδόσεις. Για τις επιδόσεις των υπηρεσιών αυτών. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής. Για να γίνει κάτι τέτοιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ανάγκη από περισσότερες πληροφορίες έτσι ώστε να μπορεί να σχηματίζει μια τεκμηριωμένη γνώμη. Οι υπηρεσίε αυτέ θα πρέπει στο μέλλον να αποστέλουν στο Κοινοβούλιο έναν πίνακα των δραστηριοτήτων του σε διετή βάση, διετή βάση. Καλό λοιπόν τις υπηρεσίες αυτές να διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους το πολιετές σε σχέση με τις κοινοτικέ στρατηγικές έτσι ώστε να βελτιωθεί γενικότερα η συνοχή. Παραδείγματα ορθής πρακτικής, βέλτιστης πρακτικής θα πρέπει να υπογραμμίζονται για να χρησιμοποιηθούν και από άλλες υπηρεσίες και αναφέρομαι σε τρία παραδείγματα. Δεν θα σας τα διαβάσω. Je vais passer à depuis le changement de statut de collège européen de μετά από την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας της υπηρεσίας, αστυνομικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ελεγκτικό συνέδριο εξέφρασε επιφυλάξεις το 2006, το 2007, το 2008 και το 2009. Εξέφρασε επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των λογαριασμών της αστυνομικής αυτής υπηρεσίας το 2007 Υπάρχουν επανειλημμένες παρατυπίες σε σχέση με τις προμήθειες, με την οργάνωση των μαθημάτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, όπως λέγεται στα ελληνικά, και η χρήση πολλαπλών και διαφορετικών κάθε φορά λογιστικών συστημάτων. Οι απαντήσεις οι οποίες έχουν δοθεί είναι μη ικανοποιητικές από πλευράς της διεύθυνσης αυτή της Ακαδημίας και σε σχέση με τα ερωτηματικά ε, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και σε σχέση με τις δικές μου ερωτήσεις και γι' αυτό εδώ σας καλώ να μην δώσουμε προσωρινά την απαλλαγή. Βέβαια από τις 16 Φεβρουαρίου υπάρχει ένας νέος διευθυντής. Οπότε ίσως να δώσουμε την δυνατότητα στην Ακαδημία αυτή να επανορθώσει τα πράγματα γρήγορα. Η επιλογή αυτή για την αναβολή της απαλλαγής μέχρι μια νέα ψηφοφορία που θα γίνει τον Οκτώβριο και η λήψη μέτρων, θυμίζω είναι από πλευρά της συγκεκριμένη υπηρεσία βέβαια, νομίζω ότι είναι κάτι με το οποίο συμφωνούν οι περισσότερες ε, πολιτικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει η Ακαδημία αυτή να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα δράση ταχύτατα σύμφωνα με τα λεγόμενα ε, στο ψήφισμα. Το πρόγραμμα δράσης αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί στις 30 Ιουνίου του 2010 και μετά έχει πολλά κεφάλαια με συγκεκριμένους στόχους που διαιρούνται σε δράσεις οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν. Για να βοηθήσουμε την προσπάθεια αυτή ζητώ από την Εσωτερική Υπηρεσία Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξουν την προσπάθεια της Αστυνομικής Ακαδημίας. Και θα πρέπει επίσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο να μας μεταφέρει τα στοιχεία που έχει για το πρόγραμμα δράσης. Για το Frontex τώρα. Η προβληματική σχετική με το Frontex έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο ως αρχή επί του προϋπολογισμού. Το ελεγκτικό συνέδριο, όπως και στις προηγούμενες περιόδους, βλέπει ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεταφορές πιστώσεων και ακυρώσεις πιστώσεων. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα πάρα πολύ σημαντικό προϋπολογισμό η υπηρεσία αυτή και οι μεταφορές ε, στην ουσία συνιστούν μια αύξηση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος. Θα ήθελα να επιμείνω στην πάρα πολύ μεγάλη σημασία που έχει μια σωστή συνεργασία ανάμεσα στο Frontex και στα κράτη-μέλη που επηρεάζουν άμεσα την εκτέλεση του προϋπολογισμού ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους. Τέλος, και για το Frontex όπως επίσης και για την Αστυνομική Ακαδημία, ο κατάλογος μελών των δικαιωτικών του Συμβουλίου δεν δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει για προφανείς λόγους διαφάνειας, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περνάω τώρα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία για τα υπόλοιπα όργανα, για τους υπόλοιπους οργανισμούς και τις κοινέ προσπάθειες, κοινέ υπηρεσίες. Γαλιλαίο, το δικαστήριο έχει, θα έλεγα, αντιμετωπίσει με σκεπτικισμό την δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με την κανονικότητα και την έλλειψη παρατυπιών. Η επιλογή της υπηρεσίας να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της χωρίς να λάβει υπόψη ότι τα προγράμματα Γκαλιλαίο και Έγνος θα μπορούσαν να διακοπούν αμφισβητείται από το ελεγκτικό συνέδριο. Από ό,τι φαίνεται όμως η υπηρεσία αυτή βρέθηκε σε μια στάση αβεβαιότητα σχετικά με τη συνέχιση των δύο αυτών προγραμμάτων, Έγνος και Γαλιλαίο. Η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνέδριου για τον Γαλιλαίο αναλύει σε μεγάλη κλίμακα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του προγράμματος Γαλιλαίο γενικότερα και κάνει συστάσεις. Τώρα για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης. Και φέτος θα πρέπει να επανέλθουμε στη διαφορά που έχει το κέντρο αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τον ορισμό του εργοδότη στα πλαίσια του καθεστώτος συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό που διαρκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ελεγκτικό συνέδριο ε, σημειώνει ότι κοστίζει πολλά εκατομμύρια στο κέντρο η έλλειψη ρύθμισης για το Eurojust. Να εκφράσω τις αμφιβολίες των συναδέλφων της Επιτροπής Λιμπέ σχετικά με τα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα του Eurojust. Δεν υπάρχουν δείκτες επιδόσεων και υπάρχουν ελλείψεις και σε επίπεδο ε, ικανοποίησης των χρηστών και σε επίπεδο ε, ισορροπίας ανάμεσα στον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εργασίας. Σημειώνω επίσης με ανησυχία ότι καμία από τις 26 συστάσεις οι οποίες ε, κυκλοφόρησαν από την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου δεν έγινε αντικείμενο εφαρμογής. Σχετικά με άλλα κοινά όργανα όπως το ΣΕΖΑΡ, ο τελικός προϋπολογισμός που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2008 δεν ήταν ιρεαλιστικός και αυτό το δείχνει το πολύ χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης των πιστώσεων. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να διαμορφώσει μια νέα λογιστική πρακτική. Το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει να παρουσιάσει μια νέα προσπάθεια έκθεσης για τον δημοσιονομικό κανονισμό που αφορά τους συγκεκριμένους αυτούς κοινούς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ο οργανισμός αυτός να έχει και εσωτερική υπηρεσία ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή standards. Και ITER, τελευταία υπηρεσία. Σας παραπέμπω στην γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Το συνέδριο διαπιστώνει ότι ο κανονισμός ITER βασίζεται στον γενικό δημοσιονομικό κανονισμό, αν και υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία απαιτούν τροποποιήσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις στην εφαρμογή των δημοσιονομικών αρχών, την καθυστέρηση στην πληρωμή των συνδρομών των μελών, όπως επίσης και άλλου είδους προβλήματα. Θα ήθελα να σημειώσω την προσοχή σας στον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου. Για τις υπηρεσίες αυτές ο δημοσιονομικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες τις οποίες έχει σε σχέση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο δημοσιονομικός κανονισμός ΙΤΕΡ δεν αναφέρεται στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ σύμφωνα με την απόφαση, με την πρόταση μάλλον του ε, ελεγκτικού συνεδρίου δεν δικαιολογείται η έλλειψη εσωτερικού ελέγχου. Θα ήθελα τέλος να συγχαρώ τρεις υπηρεσίες, ΕΦΣΟΚ, που έχει συντονίσει πάρα πολύ σωστά όλες αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες, η υπηρεσία χημικών και η υπηρεσία περιβάλλοντος. Αυτές λειτουργούν πολύ καλά. Τελείωσα. Σας ευχαριστώ κύριε Ματιού. Αναφερθήκατε σε όλα τα θέματα διαμιάς από το 21 έως το 46. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Έρενχάουζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ας επανέλθω σε αυτό που είχε μείνει προηγουμένως η κυρία Γκρέσλε σχετικά με την έλλειψη συνοχής. Βρίσκω ότι υπάρχει έλλειψη ακρίβειας. Εμείς οι ευρωβουλευτές συχνά διαμαρτυρόμαστε για το πόσο αδύναμη είναι η νομική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ φοβούμε ότι εμείς οι ίδιοι φέρουμε την ευθύνη σε ό,τι αφορά την αδυναμία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι είναι και μια ασυνέπεια που χαρακτηρίζει τις αποφάσεις μας. Ε, ζητώ συγγνώμη που πήχω. Είμαι λίγο κρυωμένος. Η έκθεση αυτή για μένα είναι απόδειξη αυτή της έλλειψης σαφήνειας. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ακριβέστεροι. Είναι σημαντικό να κάνουμε τις διατυπώσεις μας με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε να είναι μετρήσιμα τα όσα λέμε και ελέγξιμα. Έχω ορισμένε προτάσεις που μπορούν να προσθεθούν στην έκθεση αυτή. Και να πούμε και εν τέλει ξεκάθαρα ποιους οργανισμούς θα πρέπει να κλείσουμε. Για παράδειγμα, όλους τους οργανισμούς εκείνους οι οποίες με τις δραστηριότητε τους παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό το ερώτημα είναι εκρεμές από καιρό και νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι ποιοι οργανισμοί είναι αυτοί και θα έπρεπε να τους ονομάσουμε με το όνομά τους. Ταυτόχρονα να πούμε πόσα μέλη θέλουμε να έχουν τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών ώστε και εμείς να μπορούμε πλέον να ελέγξουμε και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στους οργανισμούς αυτούς. Επίσης, άλλο σημαντικό, θα πρέπει να σταματήσει η ίδρυση νέων οργανισμών εφόσον δεν έχουν πληρωθεί αυτές οι πρώτες δύο απαιτήσει τις οποίες ανέφερα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Θα ήθελε ο εκπρόσωπος μέλος του ε, ελεγκτικού συνεδρίου να πάρει το λόγο. Κυρία Αντόλοβα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Όπως γίνεται συνήθως θα λάβουμε υπόψη μας ε, τις συστάσεις σας και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την έκθεση αυτή της κυρίας Ματιό και να την ευχαριστήσω για το πολύ καλό έργο που επετέλεσε. Η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της εμπεριέχει, θα έλεγα, όλα τα σχετικά οριζόντια εγκάρσια θέματα που πρέπει να διευθετηθούν όσον αφορά την επίδοση, την χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ ότι πρέπει να στρέψουμε με ιδιαίτερη προσοχή το βλέμμα μας στις επιδόσεις των υπηρεσιών και υποστηρίζω την, ε, το αίτημα του να συντάσσονται πολιετή προγράμματα εργασίας από τις υπηρεσίες σύμφωνα με την ε, πολιετή ευρωπαϊκή στρατηγική της ΕΕ. Ένα άλλο θέμα το οποίο πολύ σωστά υπογραμμίζεται αφορά τις αδυναμίες που η ECA σε σχέση με το 2008 για τις διαδικασίες ε, αγορών αντιμετώπιση. Είναι πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες και ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρονται στην έκθεση του ECA του ελεγκτικού συνεδρίου πρέπει να αντιμετωπίσουν έγκαιρα αυτό το πρόβλημα και να υποβάλουν προτάσεις για βιώσιμες λύσεις. Επίσης η προβληματική κατάσταση του μεγάλου όγκου μεταφορών, μεταφερόμενων όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις και τις δραστηριότητες στο έγγραφο βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση. Στο τέλος εξίσου σημαντικό συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υπομειστεί τις ευθύνες της και να διαθέσει όλα, όλη την αναγκαία διοικητική ε, συνδρομή στις υπηρεσίες Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Αστυνομική Δύναμη, η κυρία Ματιό και οι συνάδελφοι οι εισηγητές γνώριζαν ότι η δική μου αρχική θέση όσον αφορά το ΣΥΠΟΛ ήταν διαφορετική. Με βάση το γεγονός ότι πρώτον υπήρξε σε σχέση με την χωρίς απαλλαγή για την ΣΥΠΟΛ το 2007 το ελεκτικό συνέδριο έδωσε συγκεκριμένη ε, θετική γνωμοδότηση για το 2008 και σύμφωνα με το ελεκτικό συνέδριο υπάρχει μια συγκεκριμένη βελτίωση της κατάστασης των πραγμάτων από το 2007 έως το 2008 ενώ όμως εκρεμούν θέματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν εγώ θεωρούσα αρχικά ότι η χορήγηση απαλλαγής θα έπρεπε να χορηγηθεί αλλά με ένα σημαντικό ψήφισμα, με ένα στεναρό ψήφισμα. Όμως είχαμε τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και τις συζητήσεις που στη συνέχεια διαμόρφωσε μια σαφή πλειοψηφία όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων για την αναβολή της χορήγησης απαλλαγής και εγώ συμφώνησα μαζί τους. Ελπίζω πράγματι ότι ο νέος διευθυντής της ΥΠΟΛ θα δραχθεί της ευκαιρία και θα αντιμετωπίσει τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ. Grazie. Se Ξαναθέλετε το λόγο, κυρία Ματιέ, για να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι. Καλώς κλείνουμε τότε. Η επόμενη συνάντηση είναι η 15η Μαρτίου. Για 10 λεπτά διακόπτομαι και στις 5.30 θα ε, συνεχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών που ξεκίνησε σήμερα το πρωί.